Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και το λόγο έχει ο κύριος Κρίστιαν Πρέντα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Προτινόμενη Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάστηκε πάρα πολύ για να στηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Οι συμβουλές μας δεν ελήφθηκαν πάντα υπόψη, άλλοτε ναι, άλλοτε όχι και τα αποτελέσματα, πώς να το πω, ε, είναι ανάμεικτα. Πώς ε, προτίθεστε να συνεχίσετε αυτή την εργασία, να εδρεωθεί θεσμικά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτίθεστε να σεβαστείτε ε, τη δέσμευση που ανέλαβε η Λέδη Άστον πριν από πέντε χρόνια να ε, είναι στο περιβάλλον της ε, κάποιος που γνωρίζει καλά και τις ευαισθησίες του Κοινοβουλίου και πότε πιστεύετε ότι θα είστε σε θέση να μας, μας φέρετε προς συζήτηση τη νέα στρατηγική που αναφέρεται στην γραπτή σας απάντηση στο ερωτηματολόγιο που σας στείλαμε. Euh, Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ε, αρχίσω να εργάζομαι για την αναθεώρηση αυτή της υπηρεσίας. Δύο πράγματα ήδη εφαρμόζονται. Άρχισα να σας το λέω προηγουμένως. Για τα υπόλοιπα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ε, εξακριβώσω τον ένδων τι ε, λειτουργεί καλά και τι όχι. Ως υπουργό είχα την ευκαιρία να το δω αυτό και μελέτησα πάρα πολύ τα θέματα. Αλλά θα με βοηθήσει η πρακτική να δω ποια είναι ακριβώς τα μέσα, οι μηχανισμοί που πρέπει να αλλάξουν ε, εκ βάθρων, ποια ε, εφαρμόζονται, έχω κάποια ε, υπόψη μου, αλλά χρειάζεται να το εξακριβώσω αυτό η δυσόμαση. Μερικά μικρά σημεία νομίζω ότι πραγματικά ε, θα πρέπει να έχουμε ε, μια καλύτερη συνεργασία ε, διαφόρων εθνικοτήτων και διαφόρων το ξέρω ότι εκπροσωπούνται κάποιες εθνικότητες ε, και επίσης συνεργασία μεταξύ εθνικών διπλωματών και υπαλλήλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ηλικιακά ενδεχομένω χρειάζεται ίσως να απλουστευτεί ε, ε, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, η αλυσίδα δίκης αν θέλετε. Θα επανέλθω σε αυτό. σε ό,τι αφορά την στρατηγική ασφαλείας νομίζω και το Απάντησα και στο ερωτηματολόγιο γραπτός ήδη. Νομίζω λέγω ότι θα είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τον Ιούνιο, του προσεχούς Ιουνίου για να τους προτείνουμε ε, κάποιες σκέψεις σχετικά με τις συστάσεις που είχαν απευθύνει το Δεκέμβριο του 2013 και ε, ενδεχομένως με αφορμή αυτό να αρχίσει μια μεγάλη δημόσια διαβούλευση και ε, προβληματισμός για το αν θα είναι στρατηγική, λευκή βίβλο, δεν ξέρω τι μορφή θα λάβει, πάντως να δούμε ποιο είναι το σενάριο αυτό των απειλών. Δύο λεπτά έχω. Καλά, τον απειλών αυτή τη στιγμή. Σταματώ εδώ, ευχαριστώ. Nein, anderthalb Minuten. ist es nur bei der S. λεπτό είχατε στη διάθεσή σας, ε, γιατί ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν ξέρω κύριε Πρέντα, θέλετε να κάνετε και μια συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, ε, κύρια Προτινόμενη Επίτροπε, θα ήθελα να μάθω αν αυτή η νέα στρατηγική θα συμπεριλαμβάνει και επανεξιολόγηση των στρατηγικών μας σχέσεων. Ε, ε, αναφερθήκατε ακροθυγώς λίγο στη Ρωσία. Δεν ξέρω, <laughs> βρήκατε τη σωστή ε, διατύπωση για να περιγράψετε τη σχέση μας με τη Ρωσία ε, για τις υπόλοιπες εταιρικέ σχέσεις. Πότε προτίθεστε να κάνετε αυτή την αξιολόγηση ή την αναθεώρηση. Ε, Μα, το θέμα και η προσπάθεια δεν είναι να βρούμε τη σωστή διατύπωση, αλλά να βρούμε τη σωστή στρατηγική και τους σωστούς εταίρους. Για το χρονισμό τώρα που με ρωτάτε, πότε θα γίνουν αυτά. Νομίζω δεν θα ήταν ε, ειλικρινές από πλευράς μου να αφαιρθώ τώρα σε ένα χρονικό ε, ορίζοντα, αλλά χρειάζεται αναθεώρηση η στρατηγική. Ο κόσμος έχει αλλάξει σήμερα. Ε, είναι τελείως διαφορετικός από τον κόσμο που είχαμε όταν κάναμε την τελευταία στρατηγική μας. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δική σας Επιτροπή νομίζω χρειάζεται να εργαστούμε από αυτόν και επί των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρωσία, προφανώς αφορά και τις υπόλοιπες. Ευχαριστώ. Ορισμένοι λένε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν μια ισχυρή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραθέτω από το ερωτηματολόγιο η Ευρώπη πρέπει να πειραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια πολιτική. Ως υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας συμμετείχατε στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών και τι μάθατε λοιπόν εκεί. Πώς μπορείτε να δώσετε καθοδηγητικό πνεύμα για να διασφαλιστεί ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πιο ενωμένοι ω προ προς τον τον κοινό στόχο. Επίσης, ε, μήπως μπορείτε να μας πείτε ένα πράγμα που σκοπεύετε να κάνετε διαφορετικά από ό,τι το έκανε η Βαρόνια Άστον. Και κάτι άλλο. Ε, πολλοί λένε ότι αν κανείς ε, θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε μία αρκούδα θα, έπρεπε, θα πρέπει να πλησιάσει αυτούς ε, που νιώθει ασφάλεια μαζί τους. Ε, γι' αυτό ρωτώ, αν εσείς έρθετε σε επαφή με μία ρώσικη αρκούδα, τι τακτική θα ακολουθήσετε. Like this committee. Μου αρέσει επιτροπή. <laughs> That's the reason why I committed myself to come. Γι' αυτό ε, πραγματικά σας λέω ότι θα έρχομαι συχνά εδώ. Λοιπόν, ε, επιτρέψτε μου να σε απαντήσω σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Κοιτάξτε, θα είμαι παρούσα, θα έρχομαι πολύ πιο συχνά, γιατί υπολογίζω στο να έχω μια ειδική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ ως βουλευτής απολαμβάνω τον κοινοβουλευτισμό. Δεν είναι καθήκον μου, είναι χαρά μου και με ενδιαφέρει και πάρα πολύ το να βρίσκομαι εδώ όσο πιο συχνά γίνεται και άτυπα και επίσημα και σε επιτροπές και σε ειδικέ επιτροπές. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε ε, θαυμάσια μαζί. Αυτή είναι η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση. Κάτι άλλο. Ως υπουργό ε, το έβρισκα πραγματικά απογοητευτικό το να δαπανά κανείς ε, ώρες ολόκληρες για το κατά πόσον η παράγραφος 2 θα έπρεπε να μετατεθεί πριν ή μετά την 6, κάτι τέτοιο δηλαδή. Ε, ώρες ολόκληρες χαλάσαμε γι' αυτό. Ξέρω ότι είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη χρήση του χρόνου σε επίπεδο υπουργών. Επίση, αν προβαίνουμε σε στρατηγικό σχεδιασμό, θεωρώ ότι έχουμε ένα θαυμάσιο δίκτυο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ανεξάντλητο πολιτικό δυναμικό και εάν λοιπόν επεξεργαστούμε μεθόδους εργασίας που θα μας επιτρέψουν όχι να ε, τρέχουμε εκ των υστέρων αλλά προληπτικά εκ των προτέρων να προβλέπουμε τι μπορεί να προκύψει. Εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω. Τώρα σχετικά με την αρκούδα δεν έχω τόσο μεγάλη εμπειρία από αρκούδες. Ίσως κάποιος από τις ε, σκανδιναβικές χώρες ε, να είναι πιο έμπειρος από εμένα. Αλλά θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε ένα μείγμα. Ένα μείγμα αυτοπεποίθησης, επιμονής και διπλωματικής, διπλωματικών ικανοτήτων. Οι αντιδράσεις θα εξαρτηθούν και από το πώς θα συμπεριφερθεί η ίδια η αρκούδα. Σε σχέση με αυτά που είπατε ε, για τη στρατηγική ε, σκέψη και το στρατηγικό σχεδιασμό, οι Υπουργοί Εξωτερικών πάντα ενδιαφέρονται για τα εθνικά συμφέροντα, κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει γι' αυτό. Το να τους πιέζει κανείς ε, να σκέπτονται στρατηγικά για να έχουμε μια καλύτερη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωστό αυτό, αλλά πώς μπορείτε να το πετύχετε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να απορρίψουμε, να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτά τα εθνικά συμφέροντα. Έχουμε κοινά συμφέροντα, γι' αυτό αλλιώ δεν θα ήμασταν μαζί. Έτσι ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώ και είναι θέμα αξιών, αλλά είναι και θέμα συμφερόντων. Φόσον λοιπόν θέλουμε και μπορούμε να μοιράσουμε αυτά τα οποία είναι κοινά, να συνεργαστούμε πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, γιατί αυτό συμφέρει όλους μας και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτύχουμε και πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Και εφόσον γίνουν όλα αυτά, νομίζω η δουλειά είναι πολύ πιο εύκολη. Δεν λέω εύκολη, πιο εύκολη. Υπάρχουν τομείς όπου βέβαια κάτι τέτοιο ενδεχομένω είναι αδύνατο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα όπου μπορούμε να επιτύχουμε πολλά αν συνεργαστούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό συμφέρον. Uh, Κύριε υποψήφια, ε, μιλήσατε για την επιθετική Ρωσία υπό τον πρόεδρο Πούτιν ε, ως βασική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Ποιος είναι ο ρόλος που σκέφτεστε για τις χώρες του κόλπου, Κατάρ και ε, Σαουδική Αραβία, για να καταπολεμήσουν τις εξτρεμιστικές ομάδες και να εξασφαλίσετε ότι η Τουρκία κάνει πραγματικές προσπάθειες για να εμποδίσει ε, τους τζιχαντιστές να περάσουν από το έδαφος της. Ε, υπάρχει συνένεση ότι το Ισλαμικό κράτος είναι απειλή. αλλά βλέπουμε ότι δεν ισχύει το ίδιο απέναντι στη Ρωσία. Ε, διαιρούμεθα απέναντι στη Ρωσία. Τι επιπλέον κυρώσει θα μπορούσατε να προτείνετε στο Συμβούλιο απέναντι στη Ρωσία, παραδείγματο χάρη να ανασταλεί η πρόσβαση της Ρωσίας στο SWIFT, ούτω ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Thank you. Uh, the... Ευχαριστώ. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας ευρύς ε, συνασπισμός ή μια ευρεία εταιρική σχέση για να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε το Ισλαμικό κράτος είναι κάτι θετικό. Και μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε εδώ στις Βρυξέλλες Ήμουν ένας από τους υπουργού ε, εξωτερικών που υπέγραψα μία επιστολή προς την ε, Λέδη Άστον στις 15 Αυγούστου, που δεν είναι φυσιολογική ημέρα για την Ιταλία και για άλλες χώρες, για να έχουμε ένα κοινό όραμα και ένα πλαίσιο για μια κοινή αντίδραση απέναντι στην απειλή του Ισλαμικού κράτους. Τότε απειλούσε μόνο ένα τμήμα του Ιράκ και φυσικά τη Συρία. Τώρα το Ισλαμικό κράτος το συζητήσαμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σε μια ευρία σύνθεση. Νομίζω ότι αυτέ οι απόπειρε είναι τμήμα τη απάντηση στο ερώτημά σα. Το να έχουμε διάφορε πτυχέ, όχι μόνο το στρατιωτικό σκέλο, αλλά να αντιμετωπίσουμε και τη χρηματοδότηση στο κίνημα, αλλά και το πολιτιστικό μήνυμα και το θρησκευτικό μήνυμα που περνάει. Τι ανθρωπιστικέ πτυχέ. Όλα αυτά είναι στοιχεία μια στρατηγική. Και το γεγονό ότι οι βασικέ χώρε που εμπλέκονται στι επιθέσει επιθέσεις είναι οι αραβικές χώρες. Και αυτή η εικόνα της γυναίκας από τα Εμμυράτα που ήταν ε, επικεφαλής ενός αεροπλάνου είναι ένα απίστευτο μήνυμα πολιτιστικά. Αυτό μπορεί να δώσει ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα στις χώρες αυτές του κόλπου. Είναι μια τεράστια κρίση, αλλά είναι και μια τεράστια ευκαιρία για τις, τους διάφορους εταίρους στην περιοχή αυτή να αρχίσουν να συνεργάζονται, γιατί υπάρχει πραγματικά κοινή απειλή, Άλλο και κοινό συμφέρον. Τώρα για την Τουρκία. Αυτό που έγινε τις τελευταίες εβδομάδες είναι απίστευτο. Ο αριθμός των προσφύγων που ελάμβανε η Τουρκία ούτως ή άλλως ήταν τεράστιος και ο, ο αριθμός των Κούρδων προσφύγων που έχει λάβει τις τελευταίες ε, εβδομάδες η Τουρκία είναι τεράστιος. Και ξέρουμε ότι τελικά ο ρόλος που μπορούμε να παίξουμε είναι να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τον διάλογο μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων της περιοχής. Για τη Ρωσία δεν έχω χρόνο μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε και συμπληρωματική 22η απάντηση όμως. Η απαντηση μας. η ομαδα μου είχε επιφυλάξεις για τη δημιουργία της ε, υπηρεσίες εξωτερικής δράσης. Τώρα όμως που δημιουργήθηκε, καταλαβαίνουμε ότι έχει αφήσει μία κληρονομιά για τις συνομιλίες της Γενέβης και, να, και για να εμποδίσουμε την αγορά πυρηνικών ε, από το Ιράν. Πώς θα βασιστείτε στην κληρονομιά της Λέδης Άστον, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε δημοσιονομική ουδετερότητα για τον προϋπολογισμό και παράλληλα να εξασφαλίσετε την προστιθέμενη δράση για τα κράτη-μέλη από την ε, δράση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. 20 δευτερόλεπτα. Θα απαντήσω καλύτερα στην ε, προηγούμενη ερώτηση. Αν η Ρωσία προσπαθήσει να πάει στο διάδρομο αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Είναι αλήθεια ότι τα κράτη-μέλη είχαν διαφορετικές ευαισθησίες για το πώς θα διαχειριστούμε την κρίση. Αλλά καταφέραμε να σταθούμε μαζί μεταξύ των κρατών μελών και των υπολείπων εταίρων μας αυτή είναι η πιο σημαντική προστιθέμενη αξία, το ότι μείναμε ενωμένοι. Και νομίζω ότι χρειάζεται να εμποδίσουμε κάτι τέτοιο από να γίνει, αντί να σκεφτόμαστε το πώς θα αντιδράσουμε αν συμβεί. Thank you very much. Κύριε Νέιτς, ευχαριστώ πολύ. Κυρία ε, Οριστήσα, είπατε πρόσωπο, εδώ είμαι. Στις απαντήσεις, στις γραπτές σας στο ερωτηματολόγιο υπογραμμίζεται την ε, ενότητα και στο στόχο και στη δράση μας για να ενισχύσουμε τη συνολική ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και της κρίσης και να μπορεί η Ένωση να γίνει όντως παγκόσμιος πρωταγωνιστής. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι αγωνίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει πάνω από μία σοβαρή κρίση ταυτόχρονα. Και όχι μόνο εμείς ε, εδώ ε, οι Ευρωπαίοι αλλά και οι περισσότεροι ε, μεγάλοι παγκόσμιοι πρωταγωνιστές. Πώς προτίθεστε λοιπόν να βελτιώσετε και να συντονίζετε καλύτερα την ανάλυση και την ε, απόκριση των διαφόρων θεσμικών οργάνων Κομισιόν, Υπηρεσία Εξωτερική δράση Συμβούλιο, Προεδρία του Συμβουλίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να τονωθεί η δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται, όχι ως αντίδραση, αλλά και ως πρόληψη καμιά φορά, αν είναι δυνατόν αυτό. Ευχαριστώ. Απάντηση, ευχαριστώ. Όπως σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή μου, πιστεύω ότι διαθέτουμε και τα εργαλεία και το πολιτικό δυναμικό. Αυτό που χρειάζεται να ενισχυθεί είναι πολιτική βούληση. Καμιά φορά αυτή έρχεται αργά γιατί αναλωνόμαστε σε συζητήσεις. Καμιά φορά έρχεται αργά γιατί αναλωνόμαστε να αποφασίσουμε. Είναι δύσκολη και ε, δύστοκη η διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Καμιά ε, ε, φορά αυτά τα πράγματα δύσκολα αλλάζουν ή είναι αδύνατα. Τα περισσότερα όμως μπορούν να αλλάξουν streamline το λένε τώρα αυτό στα αγγλικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δρομολογήσουμε με τέτοιο τρόπο τις αποφάσεις ε, ώστε να είναι πιο ορθολογική η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έχουμε πολλά εργαλεία και δυνατότητες να ανταποκρινόμαστε σε κρίσεις και υπάρχει εκεί χώρος για εξορθολογισμό. Σε ό,τι αφορά ε, την συμπροματικότητα και ε, τη συνεργασία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ανθρωπιστική βοήθεια, αναπτυξιακή βοήθεια και άλλοι τομείς πολιτικής που καταρχήν δεν έχουν σχέση με αυτά ή με τις κρίσεις, αλλά μπορούν να προλαμβάνουν κρίσεις, νομίζω ότι έχουμε μέσα ενίσχυση δημοκρατίας ή ακόμα και του εμπορίου. Γι' αυτό χρειάζεται και συντονισμό σε επίπεδο επιτρόπων για να συνδυτοποιούμε ότι είναι αλληλένδετες όλες οι πολιτικές μας. Ουσιαστικά τελικά μία πολιτική είναι εκείνη που θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να ακούγεται ε, κάπως μετέωρο ή εθεροβάμων. Θα πρέπει να έχουμε μια συνολική θεώρηση, ένα όραμα, όχι επιμέρους κάθε φορά να εξετάζουμε ένα εργαλείο, τι μας ε, χρησιμεύει, όχι. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τι θέλουμε και μετά θα βρούμε τα εργαλεία, θα τα συνδυάσουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τη σωστή πολιτική. Ευχαριστώ. Ja, guten Abend, äh, Καλησπέρα σας. Ε, μόνοι σας το είπατε ήδη. Την τελευταία φορά που είχατε έρθει είχατε πει ότι η Ρωσία δεν είναι πλέον στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το χαιρέτησαν αρκετοί για μένα και για τη δική μου την πολιτική ομάδα. Από αυτή την τοποθέτηση απορρέουν ορισμένες πρακτικής φύσεως ερωτήσεις. Δηλαδή η Ρωσία σε επίπεδο διεθνές πώς θα τοποθετηθεί σε θέματα αφοπλισμού και πυρηνικού αφοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, και του Arms Τι θα κάνει ακριβώς εκεί η Ρωσία. Πώς θα δεσμευτεί και πώς ακριβώς ε, σκέφτεστε εσείς ε, να δεσμεύσετε τη Ρωσία στη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο δημοκρατική δομή. Επίσης, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει μια νέα ειρηνική παγκόσμια δομή που να αφορά και τη Ρωσία. Και στην περίπτωση αυτή κάτι τέτοιο θα σημαίνει όχι μόνο ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, αλλά του ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που επιτρέπουν ακριβώς αυτή τη συμπόρευση. ο αφοπλισμός και ο έλεγχος των εξοπλισμών και η μη διάδοσή τους, για μένα αυτά είναι θέματα καθοριστικής σημασίας. Ως μέλος του Κοινοβουλίου έχω εργαστεί ε, Επ' αυτού επίσης ήμουν από εκείνους που υπέγραψαν αυτό το νόμο το σχετικό και η Ιταλία είναι ένα από τα πρώτα κράτη που υπέγραψε. Έχω λοιπόν κάποια γνώση και θέλω να σας πω ότι προτίθεμαι να εργαστώ σκληρά για τον αφοπλισμό, τη μη διάδοση των όπλων και τον έλεγχο των εξοπλισμών. Αυτά τα θέματα είναι συνδεμένα μεταξύ τους. Επίσης ε, προτίθεμαι ε, να μεταβώ στη Νέα Υόρκη στην επόμενη συνεδρίαση για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών NPT. Όλα αυτά είναι θέματα ασφάλειας, δεν είναι θέματα ιδεολογίας, γιατί αν κανείς εργάζεται σοβαρά για θέματα αφοπλισμού και μη διάδοση όπλων, προφανώς ο κόσμος θα γίνει πολύ πιο ασφαλής. Όσον αφορά τη Ρωσία, η Ρωσία δεν έχει υπογράψει τη σχετική συνθήκη μη διάδοση των ποινικών όπλων και θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πείσουμε τη Ρωσία να έρθει και πάλι πιο κοντά μας. Ο πρόεδρος Ομπάμα στη στην ομιλία του την προηγούμενη εβδομάδα στη... ή κάποιο, λίγο πριν από λίγο καιρό στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τοποθετήθηκε επί του θέματος και νομίζω ότι είναι σημαντικό και εμείς να θελήσουμε να φέρουμε πιο κοντά μας τη Ρωσία σε αυτά τα θέματα για τη δική μας ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο Ασφαλής, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή θέση και εγώ θα το έβρισκα καταπληκτικό <laughs> αν μετά από πέντε χρόνια είχαμε κοινή θέση. Με πολύ χαρά να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση, όσο δύσκολο και αν φαίνεται. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα όπου οι πολίτες μας ε, μερικές φορές ε, διερωτώνται και ρωτάνε ευθέως, δεν προτίθεστε να προχωρήσετε από αυτού. Έχω ξεπεράσει το χρόνο μου και γι' αυτό δεν θέλω να κάνω συμπληρωματική ερώτηση κυρία Μογκερίνη, στην Ευρώπη, λόγω του ότι υπάρχουν ένοπλες σειράξεις, σε εκατομμύρια άνθρωποι από το Ιράκ, τη Συρία, τη Γάζα και τη Λιβύη είναι πρόσφυγες. Χιλιάδες προσφύγων προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη και χάνουν τη ζωή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να ενισχύσει τους ελέγχους ε, στα σύνορα και σας ερωτώ, πώς μπορείτε να διασφαλίσετε οι συνοριακές αποστολές συμπεριλαμβανομένες και αυτή στη Λιβύη δεν θα εμποδίζουν ανθρώπους να εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να ζητούν άσυλο. Υπάρχουν αντιδράσεις στις ένοπλες σειράξεις και ο αγώνας κατά των τρομοκρατών ε, περιλαμβάνουν όλο και περισσότερο στρατιωτικές επεμβάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει ένα ψήφισμα για τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και αυτό σε σχέση με τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς θα προσπαθήσετε να θεσπίσετε ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένους στόχους. Σα ευχαριστώ. Όσον αφορά τους ετούντες άσυλο και τους μετανάστες, Είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι στις 3 Οκτωβρίου επισκέφτηκα τη Λαμπεντούζα ένα χρόνο μετά την πολύ γνωστή τραγωδία που διαδραματίστηκε εκεί. Για μένα λοιπόν είναι απόλυτα σαφές ότι έχουμε ανθρωπιστικό και ηθικό καθήκον πριν από το πολιτικό ή το θεσμικό. Το καθήκον μας είναι να προστατεύουμε τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η Ευρώπη, αυτές είναι οι αξίες μας. Βεβαίω και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το πετύχουμε αυτό, υπάρχουν πολλοί αποτελεσματικοί τρόποι. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε μέχρι άνθρωποι να διασχίζουν τη θάλασσα μπορούμε να παρεμβούμε στις χώρες προέλευσης, να προλαβαίνουμε τις κρίσεις, να επιφέρουμε σταθερότητα, να προλαβαίνουμε ενδεχομένως και δικτατορικά καθεστώτα. Μπορούμε επίσης να προστατεύσουμε τους ανθρώπους ε, που διαφεύγουν σε διάφορες ε, χώρες διαμετακόμισης, βεβαίως ε, με το σύστημα των ΗΕ και με την ύπατη αρμοστία προσφύγων, νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για τέτοιου είδους θέματα. Αυτό που επίσης πρέπει να κάνουμε είναι να λύνουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους. Λιβύη, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να επανέλθουμε αν κάποιος ρωτήσει αργότερα από αυτού. Είναι σαφές ότι είναι αδύνατον να επεξεργαστεί κανείς ένα είδος διαδρόμου αν δεν υπάρχει σταθερό κράτος. Όσον αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Θέλω να σας πω, έχω διαβάσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι ακριβώς όπως και σε όλα τα άλλα εργαλεία που υπάρχουν, τα μέσα, αυτό που τελικά είναι η ειδοποιώς διαφορά είναι ο τρόπος με, τον οποίο τα χρησιμοποιεί κανείς. Δεν είναι ναι, καλά ή κακά. Η πολιτική που εφαρμόζει κανείς κατά τη χρήση τους, αυτή είναι που ε, είναι η ειδοποιός αυτη ειναι που ειναι η ειδοποιώς διαφορα στο θέμα. Συμπληρωματική ερώτηση. <clears throat> Σε πάρα πολλούς πολέμους και κρίσεις βλέπουμε ότι διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και στη γειτονιά μας. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει κανείς ε, να τοποθετηθεί από αυτόν, να ζητήσει από τους ε, υπέτειους να, να είναι υπόλογοι. Εσείς πώς προτίθετε να το κάνετε αυτό, πώς προτίθεστε να ζητήσετε ευθύνε από τους διαπράττοντες εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, στον ε, ιστορικό αν θέλετε ρόλο που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που υπάρχει, που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το θεσμό γιατί είναι αποτελεσματικός. Αυτό ε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Thank Ευχαριστώ. Κύριε Υπάτη εκπρόσωπε, σε μία συνέντευξη 23 Μαρτίου που υπάρχει και στο blog σας, μετά την κατοχή της Κρυμαίας, εσείς δεχθήκατε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή ευθύνη γιατί είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολιτική κοινή στάση. Ακόμα και στην Ουκρανία φτάσαμε αργά. Δεν μπόρεσαμε να δράσουμε μαζί και να συλλάβουμε το εύρο τη κρίση. Αν το είχαμε κάνει του προηγούμενου μήνε, αν είχαμε προσπαθήσει την συμφωνία να την καταστήσουμε συμβατή με την ε, τελωνιακή σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όμως τους τελευταίους μήνες έχετε ε, κάπως σκληρήν τη στάση σας όταν μιλήσατε για το πώς η Ρωσία δεν είναι πια στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούν οι Ευρωπαίοι ε, γεωργοί λόγω των ε, τεράστιων απολειών που έχουν οι Ευρωπαίοι ε, γεωργοί 100 ε, εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζω η Ευρώπη να ξαναγίνει στρατηγικός εταίρος, είπατε. Πώς ε, πρέπει όμως να πορευτεί η Ευρώπη προκειμένου να γίνει πραγματικότητα αυτό. Ευχαριστώ. Το Μάρτιο έκανα αυτή την ε, συνέντευξη, είπατε. Και από το Μάρτιο μέχρι σήμερα έγιναν πολλά πράγματα, άλλαξαν πολλά πράγματα. Και μάλιστα επιταχύρω. Η Ρωσία είχε πολλές ε, ευκαιρίες για να βρει μια πολιτική ή διπλωματική λύση. Είχαμε διάφορες επαφές σε διάφορους σχηματισμούς. Ελπίζω ότι τελικά με την υπογραφή του πρωτοκόλου του ΜΙΣΚ θα έχουμε μια ευκαιρία. Και ελπίζω να εφαρμοστεί και να γίνει σεβαστό 100%. Να υπάρξει πλήρης απόσυρση όλου του στρατιωτικού προσωπικού ε, της Ρωσίας που βρίσκεται στην Ουκρανία και να υπάρξει και έλεγχος των ε, συνόρων. Για τη συμφωνία σύνδεσης, στην πραγματικότητα είπα κάτι που είναι κοινοτοπία. Ζητώ συγγνώμη. Δηλαδή, ο διάλογος ο οποίος γίνεται τώρα, ο τριμερής διάλογος, ελπίζω να χρησιμεύσει για να μειώσει τις εντάσεις. Και ούτω ώστε η συμφωνία να παίξει κάποιο ρόλο θετικό πάνω απ' όλα για την Ουκρανία και για την Ευρώπη εν συνεχεία. Ίσως για να έχει γίνει όμως αυτό καλύτερα θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει πριν. Και τώρα το κάνουμε και τώρα είναι χρήσιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είχα πει ότι καλό ήταν να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, το συμμερίζονται πολύ δεν νομίζω ότι είναι και καμιά αποκάλυψη, είναι κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό αν το πει κανεί. Το να είχαμε μιλήσει προηγουμένω ίσω θα είχε βοηθήσει. σω και όχι βέβαια, γιατί και για άλλα πράγματα ορθώσαμε το ανάστημά μα, μιλήσαμε και δεν χρησιμεύσε. Πάντω, έστω και τώρα είναι χρήσιμο να μιλήσουμε. Yes, thanks. Ε, volevo chiederle, il ritorno Το να υπάρξει ξανά εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Είναι εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση για να ξαναρχίσουμε το διάλογο με τη Ρωσία και να κυρώσουμε τις ε, κυρώσεις. Εγώ φαντάζομαι ότι πολύ δύσκολα θα εγκαταλείψει την Κρυμαία η Ρωσία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και όπως είπατε στις 23 Μαρτίου, πώς σκοπεύετε να δράσετε τούτο ώστε να μην φτάσουν ξανά στο μέλλον τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αντίστοιχα προβλήματα. Νομίζω το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό πάντα. Αυτό είναι το σημείο αφετηρία. Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση από εκεί πρέπει να ξεκινάει πάντα. Είναι αλήθεια όντω, ότι όλα όσα πρέπει να κάνουμε για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, όπως και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, θα πρέπει να αποφασιστούν κυρίω από του ανθρώπου, από το λαό τη Ουκρανίας. Ο πρόεδρο Προσέγκο επίση θα πρέπει βεβαίω να εμπλακεί μια και εξελέγει πρόεδρο πριν από λίγου μήνε ε, με καλή συμμετοχή στι εκλογέ είναι μια φιγούρα πολύ κεντρική στην όλη αυτή διαδικασία. Νομίζω κάτι άλλο με ρωτήσατε, το ξέχασα όμω. Κυρία Προτινόμενη Επίτροπε, είπατε ότι θέλετε να διασφαλίζετε την ε, ε, σύμπλευση όλων για θέματα ασφάλειας. Πάρα πολύ καλά. Και θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ο αρμόδιος ε, για θέματα τρομοκρατίας μας είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος από τους 3.000 μουσουλμάνους οι οποίοι προτίθενται να έρθουν σε ευρωπαϊκά κράτη. Αυτή λοιπόν η επιστροφή αυτών των μαχητών είναι κάτι που το φοβούνται οι αστυνομικέ αρχές όλων των κρατών μελών και διότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων. Άρα δηλαδή υπάρχουν προβλήματα και σε σχέση με τα στοιχεία τα προσωπικά, τα PNR. Θα πρέπει κανείς όλα αυτά να τα αντιμετωπίζει, αντιμετωπίζει με ρεαλισμό, γιατί αυτή η πρόκληση συνεπάγεται πολλούς κινδύνους. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω στην κυρία που ήταν ε, υπουργό η περίπτωση του Φιουμιτσίνου και η αποβίβαση στις Ιταλικές όχθες, ε, στις Ιταλικές ακτές που δεν ελέγχονται από τις ε, Ιταλικές αρχές. Και αυτό θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό και δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το μετωπίζει μόνη της η Ιταλία. Κοιτάξτε, είμαι ακόμα υπουργό Εξωτερικών της ε, Ιταλίας και σκοπεύω να παραμείνω μέχρι να αναλάβω το μου αξίωμα, όμως δεν είμαι υπουργό εσωτερικών, είμαι υπουργό εξωτερικών. Θα απαντήσω, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, οι ξένοι, οι αλλοδαποί μαχητές. Αυτό το θέμα, ε, σε αυτό πρέπει να επιδείξουμε προληπτική διάθεση. Γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε για να εμποδίσουμε την επιστροφή τους. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Και το πρόβλημα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένες ε, σταθερές ε, κατηγορίες. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο ευέλικτοι, παραδείγματο χάνει οι Υπουργοί Εξωτερικών να συνεργαστούν με τους Υπουργού Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης για να προλάβουν καταρχήν αυτό το πρόβλημα. Και σας είπα ότι είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ σύντομα συμπληρωματική ερώτηση, αλλά ο κύριος Μπροκ μιλάει δυστυχώς εκτός μικροφώνου. Περνάει στον επόμενο μιλητή, στην κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία, ε, οριστήσα είπατε εκπρόσωπο. Αντί για την ασφαλή γειτονία, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, έχουμε ε, σύνορα που φλέγονται αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση ε, χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση, όσο και έγκαιρη αντιμετώπιση των απειλών. Εσείς πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση αυτή και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς τα βλέπετε στα πλαίσια της ΕΠΑ, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και ε, στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων και των δυνατοντήτων τους. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε πολλά μέσα, πολλές δυνατότητες και πολλά εργαλεία μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και δεν τα έχουμε απαραίτητο χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, ούτε αξιοποιήσει. Είναι γεγονός ότι ακριβώς δεν φλέγονται τα σύνορα, όπως είπατε, στο παρελθόν. Είναι προφανές για μένα και ξεκάθαρο θα πρέπει να συνεργαστώ με διάφορους ενεχομένους για την προσπάθεια αυτή, αλλά για να απτύξουμε την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι προτεραιότητα. Δεν θα έλεγα υπαριθμόν γιατί έχω πολλές υπαριθμόν προτεραιότητες, αλλά είναι ε, στην ε, κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Θα πρέπει επίσης πάντα να συνεργαζόμαστε για την άμυνα, ε, χρησιμοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε τον Νοέμβριο με τους Υπουργούς Αμήνης. Ε, νομίζω θα είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που θα προεδρεύσω και θα πρέπει να το κοιτάξουμε και από την πλευρά της άμυνας, όχι μόνο για λόγους δημοσιονομικούς, αλλά και για στρατηγικούς λόγους. Χρειάζεται καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συνεργασίας. Ε, συμπροματική ερώτηση. Πώς φαντάζεστε το ρόλο του ΝΑΤΟ εκεί και εντός του ΝΑΤΟ το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενίσχυση της δικής μας κοινής ασφάλειας. Όπως σας είπα, Ήμασταν και συνάδελφοι στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και θα το γνωρίζετε από εκείνους τους καιρούς. Πιστεύω ότι η συνεργασία για την ασφάλεια με το ΝΑΤΟ είναι στρατηγική σημασία. Ήδη έχω προγραμματίσει άτυπα, γιατί εσείς θα λάβετε την απόφαση σε λίγες εβδομάδες, ε, με τον ε, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να συναντηθώ, τον κύριο Γιάννη Στόλτεμπεργκ, την πρώτη εβδομάδα ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων. Είναι διαφορετικό το σχήμα, διαφορετικές οι δυνατότητες που έχουμε, ε, διαφορετικός καν και ο αμυντικός προϋπολογισμός, ε, ακόμα και οι προσεγγίσεις καμιά φορά, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συνεργαζόμαστε με τον ΝΑΤΟ. Όταν γίνεται λόγος για τη συνολική προσέγγιση, υπάρχει και με τους εταίρους μας ε, αυτή η διάσταση συμπεριλαμβανομένου και του ΝΑΤΟ. Um, um, Ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω για τη συνεκτικότητα με την ε, ε, αναπτυξιακή πολιτική. Μιλήσατε για το συντονιστικό ρόλο στην Κομισιόν. Πώς θα δουλέψετε αυτό στην πράξη. Πώς θα δουλέψετε με τον Επίτροπο για την αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια. Πώς θα φτιάξετε προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι λαμβάνουμε υπόψη τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς θα μιλήσουμε με μία φωνή, με συνεκτικό τρόπο ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία από τις ερωτήσεις που μάλλον θα έπρεπε να απαντήσω μετά από μερικούς μήνες. Πώς θα τα καταφέρουμε. Η πρόθεση υπάρχει. Και το θετικό είναι ότι καταλαβαίνω ότι όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι επίτροποι συμμερίζονται αυτό το όραμα. Δεν θέλουν να είναι καθήκον. Όχι ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί κάποιο το αποφασίζει, αλλά υπάρχει μια αίσθηση του κατεπήγοντος. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα γύρω μας, ε, κατεπήγοντα καταστάσεις. Είτε θα συνεργαστούμε με τα διάφορα εργαλεία που έχουμε ή αλλιώς θα, θα αποτύχουμε. Ο καθένας θα αποτύχει στο δικό του τομέα, στη δική του πολιτική. Και αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο των πολιτικών μας και των εργαλείων που έχουμε. Σκεφτείτε τον έμπολα. Έχουμε αρκετά λεφτά, ξέρουμε τι χρειάζεται να γίνει, έχουμε διάφορους φορείς που κάνουν ο καθένας τα δικά του, χρειαζόμαστε ένα συντονιστικό κέντρο για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται αυτά που χρειάζονται, όταν χρειάζονται, με τον τρόπο που τα χρειάζεται ο κόσμος. Μερικές φορές χρειάζεται κανείς ένα κέντρο για να συντονίσει τα πάντα. Yes, you mentioned Ebola. And that's... Αναφέρατε τον Ebola. Πώς βλέπετε τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής, πώς θα εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια. Έχετε κάποια ιδέα για τις προτεραιότητες. Ποιο είναι το μέλλον των σχέσεων με την Αφρική. Πώς θεωρείτε θα εξελιχθεί η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Η Αφρική θα πρέπει να θεωρείται από εμά όχι μόνο ως πρόβλημα, αλλά έχει και ένα τεράστιο δυναμικό αυτή η πυρος για τη δημοκρατία, λόγω του πληθυσμού της, στην οικονομία, στην ενέργεια, το περιβάλλον. Ανάπτυξη. Ανθρώπινη ανάπτυξη. Θεωρώ ότι η Αφρική είναι τέρος. Δεν είναι μόνο αποδέκτης της βοήθειάς μας ή του ενθουσιασμού μας ή των προσπαθειών μας, ανάλογα πώς το βλέπουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε μαζί με την Αφρική, παρά να δουλέψουμε στην Αφρική. Ο κύριος Μπέντ ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Μογκερίνη. Στα νέα σας καθήκοντα έχετε και το συντονισμό και την συνοχή με άλλους τομείς πολιτικής, όπως είναι η εμπορική πολιτική. Έχω την εξής τρισχυδή ερώτηση. Πώς θέλετε να εξασφαλίσετε ε, τη συνοχή, ιδιαίτερα βάσει το άρθρο 21 της συνθήκης, στην εμπορική πολιτική αναφέρομαι. Δεύτερον, είστε διατεθειμένοι να αποσύρετε εμπορικές προτιμήσεις όταν υπάρχουν μεγάλες επιθέσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και πρότυπα. Και τρίτον, πώς θέλετε να εξασφαλίσετε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρακολουθεί και να συνοδεύει ε, ισχυρότερα την εφαρμογή και την υλοποίηση των εμπορικών συμφωνιών. Yes, thank ε, ευχαριστώ. Αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου όντως χρειάζεται να συνεργαστούμε περισσότερο. Όχι μόνο με την ε, προτινόμενη επίτροπο την κυρία Σεσίλια Μάλστρομ, αλλά και με την επιτροπή σας. Ε, ιδιαίτερα έχουμε στρατηγικές ε, συνεργασίες και όχι μόνο εμπορικές, όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική, αλλά και για πολλά και διάφορα άλλα θέματα. Δηλαδή, στο Συμβόλιο των Επιτρόπων ε, μάλλον στο σώμα των επιτρόπων θα πρέπει να συζητούμε περισσότερο και να συντονιζόμαστε. Και υπάρχει και η διάσταση αυτή που αναφέρατε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα είναι και αρμοδιότητα κάποιων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών που θα πρέπει να συνεργαστούμε και με ε, τον ΟΗΕ και βεβαίως τους υπόλοιπους αρμοδίους επιτρόπους. Για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, σας είπα, θα χρειαστώ λίγες εβδομάδες, 100 ημέρες. Νομίζω είναι ε, λογικό για να εκτιμήσω ε, πραγματικά ε, πώς λειτουργεί από μέσα αυτή η υπηρεσία, τι πρέπει και μπορεί να αναθεωρηθεί στο μέλλον πιο μακροπρόθεσμα, πιο βραχυπρόθεσμα. Τώρα δεν μπορώ να σας δώσω πιο συγκεκριμένες αποφάσεις για να είμαι απόλυτος ειλικρινής μαζί σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα αυτές που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, ε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αν θα σας απαντήσω, αυτό θα είναι από την ίδια μου εμπειρία ως υπουργό Εξωτερικών ή από τις συμπιώσει που έλαβα για την προετοιμασία μου και δεν θα ήταν ε, ε, σωστό και δίκαιο ούτε αρκετό να απαντήσω έτσι. Ωραία. Ακολουθούν κανονικές ερωτήσεις, ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση των υπόλοιπων βουλευτών από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το λίγο έχει ο κύριος Αρνό Ντανζά. Κυρία ε, Προτινόμενη Επίτροπε, ε, μιλήσατε για την αμυντική πολιτική η οποία στα τελευταία πέντε χρόνια μάλλον ήταν απούσα για να μην πω, ήταν, δεν ήταν σαφής προτεραιότητα παρά το στρατηγικό πλαίσιο που είναι φλέγον, παρά τις δημοσιονομικές περικοπές από τις οποίες πλήττονται όλοι οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Βεβαίως είναι γεγονός ότι αυτή η ευθύνη επιβαρύνει κυρίως τα κράτη-μέλη, αλλά εσείς μπορείτε να παίξετε ρόλο για να προσανατολίσετε τη συζήτηση για να λάβετε πρωτοβουλίες. Είναι σημαντικό. Εσείς πιστεύετε και εσείς, όπως καμιά φορά πιστεύει κανείς για λόγους εύκολης ιδεολογίας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιορίζεται συστηματικά σε πολιτικές αποστολές, απεμπολώντας ε, κάθε ρόλο στρατιωτικό σε άλλες συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ ή άλλα σχήματα και να περιορίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε σε μια ε, υπερ κυβερνητική οργάνωση χωρίς στρατιωτικό ε, βραχιώνα ή θεωρείτε ότι έχει ένα ρόλο να διδραματίσει εκεί. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και στις συνθήκες. Έχει ρόλο να παίξει σε αυτόν τον τομέα. Δεν τον έχει παίξει ακόμα. Θα ήταν καλό να το δούμε αυτό. Από τις ενδείξεις που είχαμε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό προκύπτει. Και θα είναι και η δική μου δουλειά να δώσω συνέχεια σε αυτή την απόφαση. Το Συμβούλιο του 2013 αποφάσισε κάτι τέτοια τον Ιούνιο θα έχουμε την ευκαιρία να προβληματιστούμε και να αξιολογήσουμε και να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πώς θα παντρέψουμε τις αμυντικές δραστηριότητες με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Κομισιόν. Μιλάω και για τον πολιτικό και το στρατιωτικό τομέα. Έχουμε ούτως ή άλλως στρατιωτικές αποστολές. Από την εμπειρία μου ε, θεωρώ ότι οι στρατιωτικές αποστολές πάνε μια χαρά, παρότι είναι περιορισμένες. Τώρα, το πώς θα επεκταθούν εξαρτάται και από την πολιτική βούληση, βέβαια. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Την πολιτική βούληση ποιών, των κρατών μελών, βέβαια. Θα πρέπει να το ξαναδούμε πάντως αυτό το θέμα. Σας είπα ότι εγώ ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας, θα, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, θα παίξω το ρόλο μου και θα συνεργαστώ με τους Υπουργούς Άμυνας, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους εταίρους μας, το ΝΑΤΟ αλλά όχι μόνο. Γιατί υπάρχει ένα δυναμικό στη συνθήκη της Λισαβόνας που δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί. Και θα προσπαθήσω τα επόμενα πέντε χρόνια να δω αν υπάρχουν οι πολιτικές συνθήκες για να το αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Ο κύριος Σάρους Βόλσκι από το ΕΛΚ. Κυρία Μοργκερίνη, η ερώτηση είναι η εξής. Πώς ακριβώς προτίθεστε να αναχαιτήσετε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αν δεν εφαρμόσετε κυρώσεις εναντίον, έναντι της Ρωσίας και αν δεν πουλήσετε όπλα στην Ουκρανία, αν δεν κάνετε και τα δύο. Από ό,τι φαίνεται η διπλωματία δεν δουλεύει, δεν θέλουμε να υπάρχει στρατιωτική σύγκρουση, δεν υπάρχει και κυρία, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Η συμφωνία του Μίνσκ ε, θεωρείται ότι πλέον δεν μπορεί και αυτή να εφαρμοστεί. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ πώς ακριβώς προτίθεστε να μας Προετοιμάστε για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Προηγουμένως είπατε ότι κάπως θα τα αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματα. Όμως η ε, στρατηγικοί και έτσι εσείς πρέπει να είστε ένας από αυτούς ε, ασχολούνται με τα σενάρια της χειρότερης περίπτωσης. Και θεωρείτε ότι η πολιτική προσανατολάς είναι ένα από τα ατού σας που διαθέτεται. Κοιτάξτε, ε, δεν ξέρω εάν απάντησα προηγουμένω, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να εργαστούμε καθημερινά με, τους, ε, με τις Ουκρανικές αρχές, με τον πρώτο Ποροσέγκο και αυτό για να μπορέσουμε να επιτύχουμε να λειτουργήσουν οι δικές του οι προσπάθειες, οι διπλωματικές και του διαλόγου. Οι προσπάθειες λοιπόν του Πρόεδρου της Ουκρανίας και του νέου ε, κοινοβούλου, γιατί θα υπάρξουν εκλογές μετά από λίγες εβδομάδες, αυτός νομίζω ότι είναι ο ρόλος μας. Να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο δυνατό σενάριο και αυτό πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε σε διάφορα επίπεδα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό έχει καμία σχέση με ε, στρατιωτική επέμβαση. Ακόμα και στην συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ότι δεν θα υπάρξει κανός είδους στρατιωτική επέμβαση και αυτό το είπαν οι ίδιοι Ουκρανοί και πρέπει να τους ακούμε γιατί σε αυτούς ανήκει η χώρα τους και σε αυτούς πρέπει να ανήκει η χώρα τους. Έτσι λοιπόν εμείς τουλάχιστον πρέπει να τους επιτρέπουμε αυτοί να οδηγήσουν τη χώρα τους έξω από την κρίση. Όμως Σίγουρα πρέπει να δράσουμε ταχύτατα ίσως ε, και να εφαρμόσουμε και περισσότερες κυρώσεις, αλλά αν τα πράγματα πάνε χειρότερα τότε μπορούμε να τις χαλαρώσουμε. Και τούμπαλιν. Υπάρχει λοιπόν και πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να στηρίξουμε περισσότερο τις πολιτικές προσπάθειες της Ουκρανικής ηγεσία. Όσο δύσκολο και αν είναι. Αν όμως δεν σταθούμε στο πλευρό τους και δεν τους βοηθήσουμε, να επιτύχουν το στόχο τους παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση που υπάρχει με την προεκλογική εκστρατεία, με το χειμώνα που θα είναι εφιάλτης και πολιτικά και ενεργειακά, με τις επικείμενες ε, εκλογές. Εάν λοιπόν δεν τους στηρίξουμε, όταν εκείνοι λένε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία πολιτική λύση, εάν δεν το κάνουμε εμείς, τότε ποιος θα το κάνει αυτό. Μαρία Γκάμπριελ. Κύριε Πατέκ, εκπρόσωποι. Στην Νότια Ευρώπη έγινε η Αραβική Άνοιξη, αλλά τι τη διαδέχτηκε, ε, ελπίδες που διαψεύτηκαν. Στην δική μας πολιτική γειτονίας μας ε, οθεί αυτή η κατάσταση να έχουμε διαφοροποιημένη στάση χώρα. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και την περιφερειακή διάσταση, ε, ειδικά σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική και δεν θα θέλαμε οι πολιτικές εξελίξεις ε, σε μια χώρα να διακυβεύονται από την αστάθεια στη γειτονική χώρα. Έχετε ένα σχέδιο δράσης για τη σταθεροποίηση της περιοχής. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, ποιε ε, πρωτοβουλίες θα αναλάβετε στο σημερινό πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο για να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ προκλήσεις. Μία ερώτηση τώρα για την Αφρική και τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό. Τι πρόταση θα κάνετε για να δουλέψουμε μαζί με του Αφρικανού εταίρους για να καταπολεμήσουμε αυτά, αυτές τις αιστείες ριζοσπαστικοποίησης που υπάρχουν στην Αφρικανική Ήπειρο και που δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις χώρες της περιοχής πάνω απ' όλα που ήταν επιτυχής. Αυτό δεν συνέβη κατά ανάγκη. Ανέφερα την Τινησία και το Μαρόκο προηγουμένως. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο την Ένωση για τη Μεσόγειο, που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους άλλους σχηματισμούς που έχουμε. Δουλέψαμε στην κρίση για τη Λιβύη τους τελευταίους μήνες με ένα σχηματισμό πενταμερή που μας επιτρέπει στο ίδιο τραπέζι να έχουμε τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γειτονικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτέ αυτές που μοιράζονται την Μεσόγειο, τις αραβικές χώρες και τις αφρικανικές χώρες. Νομίζω ότι ο αραβικός κόσμος και η Μεσόγειος γενικότερα, έχουμε αυτές τις δυνατότητες ε, να συνεργαστούμε και να, ε, και να συνομιλήσουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε θα συνομιλήσουμε υπό αυτό το σχηματισμό για όλα. Γιατί φυσικά αν πάμε προς την Μέση Ανατολή υπάρχουν άλλοι φορείς που παίζουν, με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούμε ή όχι, δεν είναι σίγουρο, αλλά πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Όταν μιλάμε για τη Λιβύη ή για το Μαρόκο ας πούμε ή για την Τινησία, θα πρέπει να κοιτάξουμε στο νότο των χωρών αυτών. Και χρήσιμο θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς να καταλάβει ότι είναι φο εταίρος και σε αυτή την περιοχή. Και στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Και στην Αφρική βέβαια. Σταματώ εδώ την απάντησή μου και πιστεύω ότι θα έχω την ευκαιρία να πω πολύ περισσότερα σε αυτό το θέμα. Thank you. Κυρία Καλνιέτε, ευχαριστώ. Κυρία Προτινόμενη Επίτροπε, δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Μόνο 18% όλοι οι Ευρωπαίοι ε, έχουν αμυντικές ε, ε, δαπάνες. Πριν από 10 χρόνια είχαμε 30%. Έτσι είναι πιο εκτεθειμένα τα σύνορά μας σε υβριδικό πόλεμο και υπάρχουν και παγωμένες λεγόμενες σειράξεις που κινδυνεύουν να ξεπαγώσουν στο κατόφλι μας. Τι προτίθεστε να κάνετε για να ενισχύσετε την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Και η δεύτερη ερώτηση συνδέεται πάρα πολύ. Ε, χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης πώς θα μετασχηματιστούν σε πιο δημοκρατικές χώρες ε, με κράτος δικαίου απέναντι στις απόπειρες της Ρωσίας να επιβάλλει τη σοβιετική ζώνη επιρροής σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για τον προϋπολογισμό τον αμυντικό. Είναι παλιά συζήτηση αυτή που κρατάει χρόνια στα διάφορα κράτη-μέλη με διάφορους τρόπους και μορφές. Αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι ε, θα πρέπει να εργαστούμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ε, για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα, το output και όχι το input. Δηλαδή όχι τα χρήματα, το πόσα χρήματα ε, δαπανώνται εκεί δεν είναι στα δικά μας χέρια. Γι' αυτό επέμεινα εγώ στην ανάγκη να εργαστούμε περισσότερο στην αμυντική συνεργασία. Αυτό ονομάζεται pooling and sharing, δηλαδή συνένωση των δυνατοτήτων και στη συνέχεια κοινή χρήση. Για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο στρατιωτικό τομέα, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να την επιτύχουμε. Σε συνεργασία με τους Υπουργούς Αμήνης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Άμυνας ε, θα ε, μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πράξη ε, συγκεκριμένα. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις απόπειρες της Ρωσίας να έχει μια σφαίρα επιρροής απολύτως στις ε, χώρες με τις οποίες συνορεύουμε προς Ανατολάς, Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε ό,τι αφορά την πολιτισμική ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντω, οι Ρώσοι προσπαθούν να κάνουν και αυτή την απόπειρα για να δείξουν ότι η ευρωπαϊκή επιλογή είναι κακή για τους λαούς αυτών των χωρών, ο ευρωπαϊκός του προσανατολισμός. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ ε, να υποστηρίξουμε τη μετάβαση και το μετασχηματισμό σε αυτές τις χώρες με αποτελέσματα προς τους πολίτες. Αν τους αποδείξουμε όλοι μαζί ότι η ευρωπαϊκή επιλογή είναι καλό για τους πολίτες αυτών των λαών. Βλέπε Μολδαβία, επί εκλογέ, δύσκολη καιρή και Γεωργία κτλ. Ε, δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει συγκεκριμένα αυτά καλά αποτελέσματα για τον κόσμο, ε, είναι ε, και αυτό ένα κίνητρο ή ένα θέλγητρο για κάποιους ε, στην κοινωνία που ε, είναι στραμμένοι προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ. <clears throat> Επόμενος μιλητής, ε, ρωτών, ο κύριος Τσέζα. Κύριε Υπουργέ, ε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου προς την Ιταλική κυβέρνηση για το ότι επέλεξε εσάς ε, ως εκπρόσωπο της δικής μας της χώρας για να μας εκπροσωπήσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή σας έχω δει πώς δουλεύετε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, συνάδελφος, είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε, θα ε, δώσετε όλο σας το πάθος ε, και ε, επειδή είσαστε και ειδικοί επί του θέματος, είμαι σίγουρη ότι πραγματικά θα είσαστε ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τις μειονότητες, τις θρησκευτικέ στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε ότι δέχονται όλο και περισσότερες επιθέσεις. οι χριστιανοί, 200.000 στο Συρία, στο Ιράκ, και έχουν αναγκαστεί λοιπόν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους ε, και κάτω από απάνθρωπες ε, συνθήκες. Έχουν κλείσει τα σχολεία, ε, έχουν καταστραφεί τα νοσοκομεία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω, επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, εσείς τι προτίθεστε να κάνετε ως ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε για τη φιλική σας διάθεση και για την ερώτησή σας. Και μέσω ημών σας σε ευχαριστώ και για τη δουλειά που έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και θα ε, υπάρξει και στο μέλλον συνέχιση αυτής της εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πείσει στο θέμα αυτό και νομίζω και εγώ μπορώ να βασιστώ πάνω σε αυτό. Εκεί λοιπόν μπορούμε να εντάξουμε ε, τις θρησκευτικές ε, ελευθερίες, την ελευθερία λατρείας και κυρίως ε, των χριστιανών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι λοιπόν σημαντικό όπως γίνεται βέβαια και από άλλους, με πολύ μεγαλύτερο κύρος από το δικό μου, να επιμείνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα οικουμενικό δικαίωμα το ε, δικαίωμα της ε, θρησκευτικής ελευθερίας. Από την άλλη βέβαια πιστεύω ότι πρέπει πολύ συγκεκριμένα να ασχοληθούμε με τα προβλήματα αυτά στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και σε κάποιες άλλες αφρικανικές χώρες, να συνεργαστούμε και με τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συνεργασία και με αυτή τη συνεργασία θα μπορέσουμε να προλάβουμε στο μέλλον παρεμφερείς καταστάσεις. Και επειδή έχω χρόνο, επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Ένα άλλο κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε κυρίως έχοντας κατά νου το Ιράκ αλλά και άλλα μέρη του κόσμου. Θέλω να πω το εξής, η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να φτάνει σε όλες τις κοινότητες. Επ' αυτού πρέπει να συνεργαστούμε με τον αρμόδιο προτινόμενο επίτροπο για να συντονίσουμε τη δουλειά μας. Προφανώς και Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική ε, που πρέπει να περάσει και στις ε, αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών και υπάρχει και μια συγκεκριμένη πολιτική. Πώς πολύ συγκεκριμένα μπορεί κανείς να μεταφέρει αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση έγινε από τον κύριο Τσέζα. Τώρα, ε, ο πρώτος ερωτών από τους σοσιαλδημοκράτες είναι ο κύριος Παρτσέρη. Ευχαριστώ κύριε Μογκερίνη. Στο προήμιο του χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο των δράσεών της. Με αυτή τη λέξη θέλουμε να τονίσουμε την, ε, και την γλυκή υπόσταση, αλλά το βιωτικό επίπεδο και στην, ε, στο της αξιοπρέπειας όλων. Αυτό που συμβαίνει στη Μεσόγειο Νομίζω ότι μας κάνει να σκεφτόμαστε αυτά που λέει ο χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, όπου ο Γιούνκερ είπε ότι είναι σημείο θετηρίας για την άσκηση των καθηκόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι χρειάζεστε χρόνο για να διαμορφώσετε τις τάσεις σας. Αλλά μπορείτε να μας δώσετε μία ημερομηνία όπου θα συζητήσετε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για τα εξή θέματα. Την ενίσχυση του ρόλου τη ύπαρτη ε, εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την προώθηση ενό συντονισμού διαρθωτικού με όλου του επιτρόπου δεδομένου του οριζόντιου χαρακτήρα που έχουν αυτά τα θέματα. Παρακαλώ, θα ήθελα ένα σχόλιο. Ε, Ευχαριστώ. Πριν λίγους μήνες, συγγνώμη, σε λίγου μήνε θα μπορούσα να σα πω ότι είναι αυτή η προθεσμία, αλλά σε κάποια θέματα θα μπορούσα τώρα να πω κάποια πράγματα και στο μέλλον θα μπορέσω να πω πολύ περισσότερα. Καταρχά. νομίζω ότι η δουλειά του ειδικού εκπροσώπου, όπως εγώ το βλέπω, ήταν πολύ θετική. Η ενίσχυση του ρόλου του, λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Νομίζω ότι το θέμα της δουλειάς ε, πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι συμπληρωματικό της εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά είναι η βάση της εξωτερικής μας πολιτικής. Και είναι και προς το συμφέρον μας. Συχνά ακούμε διάφορα ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ σταθερότητα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά το αν ε, δουλέψουμε πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα σημαίνει ότι ποντάρουμε στη σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Επομένω, θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά οριζόντιο χαρακτήρα ε, πάνω στη, σε αυτό το θέμα. Όχι μόνο για του επιτρόπου που έχουν ε, χαρτοφυλάκια με εξωτερική διάσταση, αλλά και για αυτού που έχουν χαρτοφυλάκια με εσωτερική διάσταση. Γιατί η αξιοπιστία μα απορρέει από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό των συνόρων μα. Το να είμαστε σίγουροι ότι οι εσωτερικέ πολιτικέ, λοιπόν, που προωθούμε, ανταποκρίνονται στα πρότυπα τα οποία ζητάμε όταν πηγαίνουμε να συζητήσουμε τρίτε χώρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομίζω είναι αποτελεσματικό για την αποτελεσματική, αποτελεσματικότητα τη εργασία μα. Τώρα, κάτι άλλο να πω για τη δουλειά που πρέπει να κάνω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δουλειά που πρέπει να κάνω δεν είναι μόνο θεσμική. Πρέπει να έχουμε ένα διαρθωμένο διάλογο με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, με την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη και στι τρίτε χώρε. να δούμε ποιοι έχουν προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ μίλησα για το πρόβλημα της ελευθεροτυπίας. Εδώ οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές πρέπει να εγγύψουν επί του θέματος. Έτσι, για το θέμα της ελευθεροτυπίας. Το θέμα των γυναικών. Άλλη κατηγορία. Πολύ οξύ πρόβλημα. Στο εσωτερικό, και στο εσωτερικό μας και στο εξωτερικό. Και το να δημιουργήσω μια συμμαχία θεσμική με την κοινωνία των πολιτών. Ένα μια συστηματική εργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες, είναι η καρδιά της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής μας πολιτικής. Πασκού. Ευχαριστώ, κύριο Πάσκου. Κυρία Μογκερίνη. Πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικριθεί για την έλλειψη πολιτικής βολήσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Είναι γεγονός ότι αυτό εν μέρει οφείλεται στη διαφορετική αντίληψη που έχουν τα κράτη-μέλη περί απειλών και δεν έχουν και ενιαία ευαισθησία ε, και ανησυχία. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας κατά την άποψή σας και μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις, αν θεωρηθεί να βοηθήσει να ανακουφιστεί κάπως αυτό το πρόβλημα. Ε, ελπίζω. Ε, δεν είναι τόσο εύκολο η ερώτηση, αλλά ε, αναφέρθηκα λίγο προηγουμένως σε αυτό. Νομίζω θα ήταν λάθος μας να πιστέψουμε ότι οι απειλές που τις ε, εκλαμβάνουν ως τέτοιες κάποια κράτη-μέλη δεν αφορούν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είμαστε ένα ενιαίο σύνολο, μια κοινότητα. Όταν κάποιος θεωρεί ότι έχει απειλή, θα πρέπει οι πάντες να θεωρούν ότι απειλούνται κατά την άποψή μου. Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο και την Ανατολή και τον Νότο μας ταυτόχρονα και να σταματήσει αυτή η παράδοξη εικόνα που δίνουμε είτε το ένα ή το άλλο. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να επιλέξουμε απλούστατα γιατί τα προβλήματα έρχονται και εξ Ανατολών και εκ Νότου και θα πρέπει ε, να τα αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα. Γι' αυτό σας είπα θα προσπαθήσω ε, στην αρχή ε, να προβληματιστώ για τη στρατηγική, για το όραμα, για να καθησυχάσουμε και να εξασφαλίσουμε και τους δικούς μας αλλά και τους υπολείπους. Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει όλο και περισσότερο να είναι παράγον που θα παρέχει ασφάλεια. Αλλά έχει να κάνει αυτό όντως και με την αντίληψη που έχει ο καθένας για την απειλή. E ε, κυρία υποψήφια επίτροπε, εσείς ως Ιταλίδα κατά τους επόμενους μήνες ε, θα βρεθείτε μπροστά σε ένα επώδυνο πρόβλημα για την Ιταλία πρόκειται για τους ναυτικούς που έχουν μπλοκαριστεί στην Ινδία. Αυτό αφορά την Ιταλία, άρα αφορά και γενικά το ευρύτερο σύστημα των διεθνών σχέσεων. Πρόκειται για την ασυλία, ε, την οποία διεκδικεί όμως η Ινδία για τους δικούς της ε, στο εξωτερικό. Από το 2014 γνωρίζουμε ότι είσαστε αποφασισμένοι και επειδή θα είσαστε και αρμόδια, ε, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι διμερές. Ε, εσείς ε, στις σχέσεις με την Ινδία θεωρείτε ότι αυτό το θέμα ε, θα επηρεάσει τις σχέσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ρόλο πρέπει να διαρματίσει συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, αποφάσισα ότι θα παραμείνω υπουργό Εξωτερικών ε, της ταλίας μέχρι και την ψήφο του Κοινοβουλίου. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι όσο είμαι υπουργό κάθε μεμονωμένη ημέρα θα συνεχίσω να αναζητώ μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και από τη στιγμή βέβαια που εγώ θα αναλάβω ε, άλλο αξίωμα, τότε ε, θα πρέπει να αξιολογηθεί η δουλειά που θα έχω κάνει μέχρι τότε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένα και σε πολλά επίπεδα και στο ανώτατο επίπεδο έχει θίξει αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος το έχουμε παρουσιάσει στον κύριο Μπαρόζο, στον Άστον, στον κύριο Σούλτ και στον κύριο Μπροκ, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγες εβδομάδες αυτό το θέμα των σχέσεων με τρίτες χώρες έχει σχέση με τη δουλειά της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Καταρχήν, οι Ινδικές Αρχές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και αυτό είναι και προς το συμφέρον τους. Και όπως είπατε υπάρχουν ε, θεμελιώδεις νομικές αρχές που θα πρέπει να διαφυλάσσονται από την Ευρώπη, την Ιταλία και την Ινδία που όπως είπατε κι εσείς ε, η ίδια η Ινδία ε, θα πρέπει να θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα. Το τρίτο που θέλω να κάνω προφανώς είναι να διευκολύνω το διάλογο ανάμεσα στην Ιταλία ως μέρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μεταξύ Ιταλίας και Ινδίας. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο πρόεδρος Σούλτς και η κυρία Άστον έχουν πει κατά το παρελθόν ότι αν επιληθεί σωστά, αν έχει αίσιο τέλος αυτή η υπόθεση, σίγουρα αυτό θα βελτιώσει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία. Ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη. Στην αρχική σας παρέμβαση μιλήσατε για τη σημασία των σχέσεων ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ποιες πολιτικές ε, πρωτοβουλίες θα αναγγείλετε, ούτω ώστε να βγει από το αδιέξοδο η διαδικασία διαπραγματεύσεων για την σύναψη συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Διαδικασία η οποία έχει βαλτώσει από τη δεκαετία του 90. Καταλαβαίνετε ότι πέρα από τις οικονομικές και εμπορικές ε, διαστάσεις έχει μια τεράστια σημασία αυτό το θέμα. Ε, δίνουμε τεράστια σημασία αυτή τη στιγμή στο TTIP, τη διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Καλώ. αλλά μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εμπορικές, οικονομικές και πολιτιστικέ σχέσεις μας με τις χώρες του Μαρκοσούρ. Το ερώτημά μου είναι απλό. Τι βαθμό προτεραιότητα θα δώσετε σε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ κύριο Μπέλντερ, λέει ο πρόεδρο. Ναι, μήπως να απαντήσω πρώτα. Φεδερίκα, I so much Italian understanding, so, eh, Έχεις το λόγο. Να απαντήσω στα Ιταλικά. Σε μια λατινική γλώσσα, από όλε τι λατινικέ γλώσσε, επιλέγω τα, Ιταλικά. Πριν από δύο μήνε στο Σαντιάγκο τη Χιλή με το Γενικό Γραμματέα της ΕΛΑΚ συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Και είπα τότε, πριν από δύο μήνες, νομίζω ότι κάπου θα υπάρχουν κάποια πρακτικά αυτής της συνάντησης, ότι η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής μπορεί να γίνει ακόμα πιο ουσιαστική ακόμα πιο θεμελιώδης. Έχουμε μια κοινή βάση σε ό,τι αφορά τις πολιτιστικές, ιστορικές σχέσεις, την αμοιβαία κατανόηση, ακόμα και τις πολιτικές σχέσεις. Έχουμε δομές. Δημόσιου βίου, ας πούμε, στη, στη ζωή μας, δημόσιου βίου στη, στην Ευρώπη και στην ε, Λατινική Αμερική, κοινέ. Και κατα, καταλαβαίνουμε στον άλλον εύκολα. Αυτό που λείπει είναι μια ακόμα πολιτική δέσμευση, μια μικρή ακόμα επιπλέον πολιτική δέσμευση, αν θέλετε, ούτω ώστε αυτή η εταιρική σχέση να αναπτυχθεί 100%, να αναπτύξει όλο το δυναμικό που εμπεριέχει. Αυτό νομίζω ότι ισχύει και για το Μερκοσούρ, αλλά και για τι άλλε περιφερειακέ οργανώσει που υπάρχουν στη Λατινική Αμερική. Κάθε μία από αυτέ έχει τι δικέ της πολιτικέ αποχρώσεις. Φυσικά, το ξέρω πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να συνεργαστούμε με μεγαλύτερη όρεξη με μεγαλύτερη ζέση προς αυτό το στόχο. Όχι μόνο με τη Λατινική Αμερική, αλλά και με την Καραϊβική. Και έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Που... Έχουμε τη Σύνο Κορυφής. Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΑΚ, τον Ιούνιο. Για μια φορά μπορεί να είναι όχι το business as usual με την αρνητική χρειά, αλλά με τη θετική χρειά. Μπορεί να γίνει μια στιγμή όπου ξαναδείχνουμε την βούλησή μας να συνεργαστούμε. Όχι μόνο με τις χώρες που είναι για μας στρατηγική εταίρη, αλλά με όλη την Ήπειρο. Εμπέλα. Κύριος Μπέλτερ. Eh. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ μιλάω Ολλανδικά, κύριε Μογκερίνη. Ε, αυτό τον καιρό βλέπουμε και παγκοσμίω και περιφερειακά μια αποσταθεροποίηση από τρομοκρατικές οργανώσεις μουσουλμανικές, Χεσμπολά, Αλκάιντα, Άιζης, Χαμάς και πάει λέγοντας. Και στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παράλληλα συμφέροντα ασφαλείας. Συμφωνείτε, αν όχι γιατί και αν ναι, πώς ε, αυτό θα μεταφραστεί ε, συγκεκριμένα στην πράξη, στην πολιτική ε, ασφάλειας και άμυνας. Ευχαριστώ. Κυρία Μογκερίνη. Συμφωνώ ότι υπάρχει μείζων απειλή που προέρχεται από παντού, ολόγυρά μας. Αλλά αυτό αφορά κυρίως τους πολίτες της εκεί περιοχής κατά κύριο λόγο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτή την άποψη μαζί μου. Τα πρώτα ε, θύματα του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν και χριστιανοί και άλλοι, αλλά τα πρώτα θύματα είναι μουσουλμάνοι. Και αυτό είναι και μια θεώρηση που θα πρέπει να έχουμε. Και το πολιτιστικό μήνυμα που στέλνουμε εμείς σήμερα είναι ένα τμήμα της στρατηγικής για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Γιατί η αφήγηση που χρησιμοποιεί ε, το Ισλαμικό ε, λεγόμενο κράτος είναι ακριβώς ότι ε, αυτό αποκαλείται κράτος ενώ καταλύει την έννοια του κράτους και την καταστρέφει. Την κρατική κυριαρχία, τα σύνορα κτλ. Από την άλλη χρησιμοποιεί μια θρησκεία κατά των άλλων θρησκείων. Αυτά όμως δεν έχουν καμία βάση ούτε στο Ισλάμ ούτε σε καμία θρησκεία. Λοιπόν, το πολιτισμικό μήνυμα που θα πρέπει κυρίως να έρχεται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και ισχυρό μέσο. Έχουμε και άλλα μέσα και τα στρατιωτικά προς το παρόν. Ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να το χρησιμοποιήσουν, κάποια άλλα όχι, κάποια τρίτα με άλλο τρόπο. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που θα κάνουν στο μέλλον και πάλι, τι είναι. Να δημιουργήσουμε ένα κοινό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί να λειτουργεί προς την ίδια κατεύθυνση και να δρά. Θα υπάρχουν δυνατότητες που θα παραμείνουν στα χέρια των κρατών μελών, αλλά αν αυτές οι αποφάσεις και αυτές οι δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που τους ε, καθοδηγεί, τους δείχνει την κατεύθυνση και τη στρατηγική και συνενώνει τις δυνάμεις, τότε έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και αποφεύγουμε να αποκλίνουμε και να μιλούμε με πολλές φωνές. Και ε, μετά έχουμε την ε, ανθρωπιστική πτυχή, που είναι και τεράστιο το ζήτημα. Και μπορεί αυτό Α, συγγνώμη, τελείωσε ο χρόνος μου. Um, uh, Κυρία υποψήφια uh, επίτροπε, μιλώ εκ μέρους του κυρίου Βανόντα που δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει σήμερα και μου ζήτησε να κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, προς εσάς. Ποιες δραστηριότητες πιστεύετε ότι πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν μπορεί να τις αναλάβει το ΝΑΤΟ ή συνασπισμός κρατών. Και το δεύτερο, πιστεύετε ότι ο στόχος είναι να προαχθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πώς η Ευρώπη θα γίνει ένας παγκόσμιος παίκτη. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι αποστολές μας ε, δεν είναι ότι υπάρχουν επειδή δεν μπορεί κανείς ε, να τις αναλάβει. Εγώ πιστεύω ότι από μόνοι μας αυτό που κάνουμε είναι πολύ σωστό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτά που δεν κάνουν οι άλλοι, που μας τα αφήνουν ως κατάλοιπα, δηλαδή κάτι που δεν κάνουν τα κράτη-μέλη ή το ΝΑΤΟ. Και βεβαίως ε, υπάρχουν και αποστολές ε, και επιχειρήσεις όπου συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη και με τον ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο και σοφό να υπάρχει έτσι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ξέχασα, φοβάμαι ότι ξέχασα το δεύτερο σκέλος ερώτησή σας. Κοιτάξτε, δεν θα δαπανούσα τόσο χρόνο διερωτώμενοι γιατί, αλλά πιο πολύ χρόνο για να κάνω το σωστό. Και ο βασικός λόγος είναι ότι χρειαζόμαστε κάτι που να είναι χρήσιμο, όχι κάτι που να μας κρατάει απλά ενωμένους, κάτι που να είναι χρήσιμο για την ασφάλεια τη δική μας και των υπολείπων. Ο κύριος Ντέμες Μάκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Μόγεριν, μιλώ και εγώ Ολλανδικά. Θα ήθελα λίγο να επανέλθω στη φιλοδοξία να μπουν στο κέντρο της εξωτερικής δράσης τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εκεί. Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει η Σύμβαση των ΟΕΕ κατά των βασανιστήριων. Δυστυχώς παντού επιδεινώνεται η κατάσταση ανά τον κόσμο και σε ό,τι με αφορά νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει αυτή την κακοποίηση και τα βασανιστήρια. Εσείς θα το θέσετε αυτό ως πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ε, ένα ψήφισμα ε, για την ε, αφαίρεση οργάνων από τα μέλη της οργάνωσης Falun Gong στην Κίνα από διαφόρους ανθρώπους. Θα φροντίστε να τερματιστεί αυτό με μια έρευνα διαφανή και ελεύθερη και να φεθούν όλοι οι ελεύθεροι που κρατούνται για αυτό το λόγο. Uh, yes, I, uh, Μάλιστα. Βεβαίως με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα των βασανιστήριων, όπως και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι μόνο ύψιστη προτεραιότητα, θα είναι ένα πόσπαστο στοιχείο στον πυρήνα της δράσης μας. Βεβαίω έχουμε πολύ μεγάλη πραγματογνωμοσύνη, όχι μόνο εμεί στο εσωτερικό των υπηρεσιών, αλλά και στι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Σα είπα ότι χρειάζεται και να σφυριλατηθεί εκεί μια συμμαχία με τι οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ακτιβιστέ και την κοινωνία των πολιτών στι ίδιε τι χώρε που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και αυτό θα είναι ένα τμήμα των καθηκόντων μου, όπου μπορώ να το αναφέρω. Αλλά εκτός αυτού, κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχουμε αποφασιστική δράση που να κάνει τη διαφορά και αυτό έχει να κάνει με την Κίνα. Και θα είναι και ένα θέμα που θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τις κινέζικες αρχές. Τι προσπαθώ να κάνω εγώ. Ε, διάφορες χώρες να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια όχι να τους στιγματίζουμε, να τους λέμε τι πρέπει να κάνουν, να τους βοηθήσουμε για να αλλάξουν αυτές τις πολιτικές και αυτές τις πρακτικές. Αυτό νομίζω είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφερθήκατε στο Hong Kong στην τελευταία σας ερώτηση, ε, αν δεν σας κατάλαβα καλά. Ε, α, μήπως δεν σας κατάλαβα εγώ. Ε, Έχω λίγο χρόνο, δεν μπορώ να απαντήσω. Σήμερα, μάλλον τα νέα από εκεί είναι ευχάριστα και όχι τόσο άσχημα. Και αυτό ε, είναι ε, προς τιμή ε, όχι μόνο των αρχών του Χονγκ αλλά και της Κίνας για να λυθεί μέσω του διαλόγου το θέμα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σχάκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία είπατε, εκπρόσωπε, είπατε ε, ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε γενικά αλλά να δρούμε αποτελεσματικά. Ένα επικοδομητικός εταίρος, η Ρωσία, πώς θα το κάνουμε αυτό και πώς βλέπετε το ρόλο σας στο, στις διαπραγματεύσεις P5 συν 1 για το Ιράν ε, και πώς θα εμπλακεί και ο λαός του Ιράν εκεί για να αντιμετωπίσουμε ε, όλα αυτά τα θέματα και τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Εσείς μπορεί να είστε αισιόδοξοι, αλλά ε, μπορεί είναι μια προσπάθεια αυτή που κινδυνεύει να τραβήξει σε μάκρος και να διαονίζεται. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Είπα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Ιράν θα μπορούσε να παίξει ένα επικοδομητικό ρόλο και θα μπορούσε να παίξει όμως και ένα καταστροφικό ρόλο στην ε, περιοχή, σε διάφορες συγκρούσεις που έχουμε στην περιοχή. Γι' αυτό είναι σωστό να εμπλέξουμε το Ιράν και να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να είναι τμήμα της λύσης και όχι κάποιος που προκαλεί την καταστροφή. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό τουλάχιστον να προσπαθήσουμε, όπως κάναμε και με το Ιράκ. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τις χώρες που μπορούν να που παίζουν ένα ρόλο. Και κυρίως με, το, με τους ανθρώπους που εντός της χώρας που παίζουν ρόλο. Ε, για τις διαπραγματεύσεις B1+. Ε, οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στις 24 Νοεμβρίου. Η Λέδη Άστον θα συνεχίσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Είναι πολύ σωστή απόφαση, προφανώς δεν αλλάζουμε διαπραγματευτή τις τελευταίες εβδομάδες σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Μίλησα και με την Κάθη, αλλά και με τους άλλους εμπλεκόμενους υπουργούς, αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών της, ε, του Ιράν. Και είτε θα φτάσουμε σε συμφωνία στις 24, πριν τις 24 Νοεμβρίου, ή θα γίνει πολύ δύσκολο να συμφωνήσω μετά. Και ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δύο θέματα θα πρέπει να παραμείνουν χωριστά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπερβολικά σημαντικά για να μπερδευτούν οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση. Όπως είπα, συζητάνε το πυρηνικό φάκελο. Και πέρα από το περιφερειακό ρόλο του Ιράν, θα πρέπει πάντα να υπάρχει το θέμα, η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάντα θα πρέπει να θέτουμε αυτό το θέμα στις Ιρανικές αρχές. Ο κύριος ε, Μαούρα Μπαραντιάρα. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Οριστήσα, είπατε εκπρόσωπε, σας ερωτώ για τη διμερή σύνθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβας. Κανονικά αυτό θα πρέπει να συνδέει την ε, διάνοιξη της οικονομίας με τις ελευθερίες ε, ε, στην Ίσο. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις δεν ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα του κουβανικού λαού. Σας ερωτώ πρώτον, συμφωνείτε οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις του καστρικού καθεστώτος είναι απλώς επιπόλες και δεύτερον, Είστε διατεθειμένοι να αρχίσετε ένα επικοδομητικό διάλογο για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή με τις κουβανικές αρχές. Και αν είναι καταφατική απάντηση, πώς θα παρακολουθήσετε τη σωστή ε, ανάπτυξη των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ρόλο θα έχει εκεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εποπτεία και την επιτήρηση. Και τέλος, κυρία Μογκερίνη, σε περίπτωση που εκλεγείτε και που επιβεβαιωθείτε θα σας παρακαλούσα ε, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και οι αρχές του και αξίες του για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κυριαρχούν επί των οικονομικών συμφερόντων σε όλες τις αποφάσεις που θα λαμβάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω σίγουρα, αν μου το επιτρέπετε, αν το επιτρέψετε, αν αποφασίσετε. Θα επανέλθω λοιπόν μετά από λίγους μήνες αυτό το θέμα, αν μου το επιτρέψετε με την επιβεβαίωσή μου. Και θα σας μιλήσω για τα επόμενα βήματα, γιατί πρέπει να γίνει. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι, από τη μία είμαι πεπισμένη, ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το μικρό αυτό άνοιγμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που γίνεται από τις αρχές. Μπορούν να γίνουν περισσότερα, προφανώς, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο και κυρίως σε πολιτικό επίπεδο πιστεύω ότι ο ρόλος μας είναι να ενθαρρύνουμε και να οθήσουμε ούτω ώστε η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων να είναι πιο πλήρης, πιο πιστική και να προχωρήσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Είμαι έτοιμη βεβαίως να ξεκινήσω ένα επικοδομητικό διάλογο, όπως είπατε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κουβανικές αρχές. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω με τον ειδικό εκπρόσωπο μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα έχω τη χαρά να συνεργαστώ μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τη μορφή που εσείς κρίνετε καταλληλότερη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μορκερίνη, Χαίρομαι που δώσατε ιδιαίτερη σημασία στο να υπάρχει ε, συνέχεια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος ε, με τον οποίο καλύψατε όλες ε, τις διαστάσεις και τις κατευθύνσεις των εξωτερικών μας σχέσεων και πόλεων. Επίσης, θέλω να σας πω ότι επειδή προέρχομαι από τη βόρεια χώρα, χάρηκα πάρα πολύ για αυτά που είπατε για την Αρκτική. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς είμαστε ηγέτιδα δύναμη σε τρεις τομείς, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας σε παγκόσμια κλίμακα μέσω ε, συντονισμών και μέσω μιας συνεπούς πολιτικής. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει και να συνεργαστείτε με τους άλλους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ θα δώσω όλη μου την ενέργεια. Είναι σημαντικό να θέτει κανείς υψηπετή στόχους. Ε, επίσης, όταν ε, Πρόκειται για το εμπόριο, για το περιβάλλον. Ε, είναι δύσκολο να πει κανείς τώρα πώς ακριβώς θα συντονιστούμε. Νομίζω ότι ο συντονισμός, ίσως τώρα αυτή να είναι μια μεσογειακή προσέγγιση, παρότι η Αρκτική είναι στην καρδιά μου, είναι μια πολύ όμορφη και στρατηγική σημασία περιοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι ο συντονισμός ξεκινάει με το να μοιράζεται κανείς ιδέες, προτεραιότητες και εργαλεία. Και γι' αυτό το λόγο στις ε, μηνιαίες ε, συναντήσεις που οργανώνουμε με τους άλλους επιτρόπους και δεν αναφέρουμε μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και με άλλους που ασχολούνται με θέματα εσωτερικής πολιτικής ας πούμε για το περιβάλλον, το χρειαζόμαστε και αυτό. Και αυτούς που ασχολούνται με θέματα εμπορίου. Και αυτούς τους χρειαζόμαστε. Μόλις λοιπόν αρχίσουμε να μοιραζόμαστε τα οράματα και τα εργαλεία, τότε θα δούμε κατά πόσον ο μηχανισμός θα λειτουργεί ή όχι. Αυτή είναι η πρόκληση. Δηλαδή να δίδουμε μια, ένα πολιτικό περιεχόμενο στις ε, διάφορες δομές που υπάρχουν έτσι ώστε και οι δομές αυτές να συνεργάζονται. Αυτή είναι η πρόκληση. Τώρα σε θέματα παγκόσμιας εμβέλειας αυτό που κάνουμε στην Αϊτή ή στο κέρας της Αφρικής. Αυτά είναι τεράστια, είναι πολύ σημαντικά. Και βεβαίως προχωράμε σταδιακά και αν τελικά κατορθώσουμε να τα συντονίσουμε όλα αυτά και να τους δώσουμε μια πολιτική μορφή, προφανώς θα είναι πιο σημαντικά, πιο ορατά και γνωρίζουμε ότι η πολιτική παρουσία, το να φαίνεται κάτι, είναι πιο ισχυρό και γίνεται και πιο ελκυστικό για τους άλλους. Για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή ε, θα πρέπει να εργαστούμε από αυτού στη Λίμα και στο Παρίσι έτσι ώστε να πετύχει η όλη υπόθεση. Γιατί αν δεν πετύχει αυτό είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ οποιαδήποτε άλλη επιτυχία στο μέλλον. Ήβο Βάγγελ παρακαλώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, Όταν ήσασταν εσείς στη Λαμπεντούζα, εγώ ήμουν στην Αντίσα Μπέμπα. Και όταν ήμουν εκεί, πίστηκα ότι ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων θα αυξηθεί στο μέλλον, εάν δεν καταφέρουμε να προετοιμάσουμε διαρθρωμένες πολιτικές για την Αφρική. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αποφασίσατε να προετοιμάσετε μια τέτοια πολιτική. Είπατε επίσης ότι έχει σημασία το διεθνές δίκαιο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιήσει αυτό το δίκαιο, νομίζω ότι θα γίνουμε πιο σημαντικός ε, πέκτης και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ε, στο θέμα της, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και στο θέμα της Σαχάρας. Θα χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε όταν κάποιος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πολύ συμβολικό το ότι ήσασταν στην Αντισαμπέμπα ε, όταν εγώ ήμουν στη Λαμπεντούζα, γιατί ακριβώς αυτός είναι ένας από τους δρόμους που χρησιμοποιείτε. Αυτό που με εντυπωσίασε ακόμα περισσότερο ήταν η συνάντηση με τους συγγενείς των θυμάτων στη Λαμπεντούζα και τους ε, επιζήσαντες. Δεν με εντύπωσαν τόσο οι ιστορίε των ανθρώπων που πέθαναν, αλλά οι ιστορίε των ανθρώπων που επιβίωσαν. Είδαμε την τραγωδία στη θάλασσα, αλλά συχνά ξεχνάμε τι προηγείται πριν μπουν αυτοί σε αυτά τα σκάφη αυτοί οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Μιλάμε για βασανιστήρια, παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα παιδιά, για τι γυναίκε και για του άντρε. που στις περισσότερες περιπτώσεις για τη Λαμπεντούζα οι άνθρωποι που περνάνε από τη Λιβύη στην Ιταλία είναι κυρίως ε, ετούντες άσυλο, είναι πρόσφυγες. Δεν είναι οικονομικοί μετανάστε. Επομένω, σίγουρα χρειαζόμαστε μια ειδική πολιτική για την Αφρική. Και για το καλό τη Αφρική, αλλά και για το δικό μα το καλό. Για το διεθνέ δίκαιο. Φυσικά, αν είμαι έτοιμη να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία Φυσικά μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, αλλά πριν από αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε μια προληπτική πολιτική. Αν κοιτάξουμε όλες τις κρίσεις που έχουμε, όλες, αναφέρατε τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει αυτή η ιστορία ε, μεγάλωσα με αυτή τη σύγκρουση. Άλλες συγκρούσεις βλέπαμε ότι ετοιμάζονται και οφορούνται, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να τις παρεμποδίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να σκεφτόμαστε τις κυρώσεις μετά αφού ξεσπάσει ο πόλεμος, το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να αποτρέψουμε τις συγκρούσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόουσο Κυρία Μογκερίνη, η κατάσταση στο Ιράκ και στη Συρία είναι απόρρια των δυτικών πολιτικών των τελευταίων 20 ετών. Θα με καταλάβετε καλύτερα αν σα αποτύσσω ε, ένα μικρό φόρο τιμή στον Μπερνάρντο Μπερδοτολούτσι, ο οποίο, αν σήμερα σκηνοθετούσε το 1900 θα μα έδειχνε ότι ο ακραίο Ισλαμισμό όπω και ο φασισμό, δεν είναι σαν τα μανιτάρια που βγαίνουν ξαφνικά τη νύχτα. Οι δυτικές δυνάμεις ε, τα έσπηραν όλα αυτά, τα θέλησαν και τα πληρώνουν τώρα και με τους ε, Ισλαμιστές οι δυτικέ δυνάμεις κάθε φορά κέρδιζαν περισσότερα. Ε, μέχρι και δεν ξέρω πια τι να το κάνουν το πετρέλαιο και έτσι μας έφεραν στον πόλεμο που πληρώνουν οι ίδιοι τα σπασμένα. Οι νέοι μας και οι λαοί που θέλουν μόνο να έχουν μια ζωή αξιοπρεπή και σε ειρήνη. Το κακό ονομαζόμενο Ισλαμικό κράτος είναι απόρρια της εισβολής στο Ιράκ και τη Συρία. Και την, ε, ε από όλη την αποτυχία στη Συρία. Τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να δίνουμε περισσότερα όπλα σε αυτές τις θρησκευτικέ ε, φατρίες. Εσείς είστε προσιλωμένοι ε, στην ενότητα και την εδαφική ακαιρεότητα του Ιράκ και της Συρίας. Η εδαφική ακαιρεότητα και της Συρίας και του Ιράκ είναι θεμελιώδου σημασία. Πιστεύω όμως και κάτι άλλο, και εδώ δεν θα συμφωνήσουμε, ότι είναι εκ των όνων κάνεθ, είναι καθήκον να βοηθήσουμε και μέσω παροχής όπλων, μέσω προμήθειας όπλων, αν και αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς ανταλλάσσουμε απόψεις. Να βοηθήσουμε τους ε, όσους αντιστέκονται σε μια τρομοκρατική οργάνωση που απειλεί τη ζωή τόσων πολλών αμάχων. Είναι νομίζω ανθρωπιστικό καθήκον να το κάνουμε. Και εξάλλου δεν υπάρχει και στρατιωτική απάντηση και εδώ συμφωνούμε εάν δεν υπάρχει πρώτα πολιτική απάντηση. Και αν δεν δουλέψουμε πάνω στις συνθήκες που μας οδηγούν που μας οδηγούν στον πολλαπλασιασμό των, των εξτρεμιστών. Ε, αστάθεια, φτώχεια, κοινωνική αβεβαιότητα, οικονομική αβεβαιότητα, βαθύτατες κρίσεις, βαθύτατα χάσματα, αποκλεισμοί που δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί τη στρατολόγηση ατόμων από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό νομίζω είναι το βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και όλων μας επιμέρους να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Γιατί? Γιατί οι καλύτερες συνθήκες ζωής, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικές συνθήκες, οικονομικές συνθήκες, κοινωνικές συνθήκες στις χώρες που είναι γύρω μας, σίγουρα θα αφαιρούσε πόρους από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που απειλούν τους πληθυσμούς, από τους οποίους βρίσκουν μαχητές λόγω της απελπισίας τους. Ο κύριος Ιγκλέσιας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρία Μαγκερίνη οι δικές μου παρεμβάσεις εδώ είναι σκληρές και επικριτικές συνήθως, αλλά θα κάνω σήμερα μια εξαίρεση. Παρόλο που έχουμε τεράστιες διαφορές, θα πρέπει ο καθένας να έχει την ευκαιρία ότι μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. Σας ομολογώ ότι μερικές από τις επικρίσεις που σας έγιναν, ε, σας κατέστησαν πολύ συμπαθή στα μάτια. Σας είπαν ότι είστε ε, φίλοι των Ρώσων. Ε, που θα ήταν σαν να μου λέγανε ότι είμαι φαλακρός εγώ. Ε, είπατε, ακούστηκε ότι είστε εμπειρογνώμων χαμηλού προφίλ. Όσο και αν αγαπάτε το ΝΑΤΟ, εγώ νομίζω ότι έχετε και πολύ κοινή λογική και πάρα πολύ καλή κατάρτιση. Αυτή η κοινή λογική είναι κάτι που λείπει πολύ συχνά εδώ. Λέτε ότι θα έρχεστε με πολύ μεγάλη χαρά. περίεργε χαρέ οι δικέ σα που φαίνονται. κυρία Μογκερίνη, ο Γούντι Αν έλεγε ότι δεν μπορεί να ακούσει Βάγνερ γιατί του έρχεται να εισβάλλει στην Πολωνία. Και εδώ ορισμένοι ακούνε τόσο πολύ Βάγνερ που τους έρχεται να εισβάλλουν στη Ρωσία. Και περισσότερο από ερώτηση θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το εξής περίεργο. Ε, απαντώντας στον κύριο Καστάλτο είπατε ότι αρχές της ε, διεθνούς νομιμότητας θα πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστές. Σας ερωτώ, η τόσο πολεμοχαρής Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία δεν σας φαίνεται ότι έρχεται σε αντίφαση με την ανοχή και την ε, καλοσύνη με την οποία αντιμετωπίζουμε το Ισραήλ που τόσο συχνά παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν θα τοποθετηθώ για αυτό που είπατε για τις χαρές. Ο καθένας έχει τις δικές του χαρές. Τι να κάνουμε. <clears throat> Ομολογώ όμως ότι σε πολιτικό επίπεδο, όπως συμβαίνει εδώ, σε αυτή την αίθουσα, το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο, όχι μόνο για τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, μαζί, μόνοι μας, ο καθένας σε διαφορετικό ρόλο, αλλά το βρίσκω και πάρα πολύ σημαντικό ε, σε διανοητικό επίπεδο. Σας ομολογώ ότι για μένα αυτή η εξέταση, όπως παρουσιάζεται, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για τις ερωτήσεις που παίρνω. Γιατί πίσω από κάθε ερώτηση κρύβονται πάρα πολλές ε, απόψεις και ιδέες. Δεν θέλω να ξεφύγω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που συμμεριζόμαστε αυτή την ε, ιδιαίτερη χαρά. Τώρα, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς αρχές νομιμότητας, πράγματι ισχύουν για όλους. Και με εκπλήττει το γεγονός ότι είναι η πρώτη ερώτηση που θίγει το θέμα της Μέσης Ανατολής. Εγώ θα περίμενα περισσότερες ερωτήσεις ε, σχετικά με τη Μέση Ανατολή από εσάς σήμερα. Μπας περιπτώσει, πιστεύω ότι στη, Μέση στη Μεσόγειο το βασικό μας καθήκον είναι να ασχολούμεθα με τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο γιατί είναι ένα θέμα που αφορά το Ισραήλ και το Παλαιστίνη είναι τουλάχιστον δύο συγκρούσεις είναι οι αραβικές χώρες και το Ισραήλ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι και η πιο σωστή προσέγγιση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εκεχηρία που επιτέχθηκε με πολύ μεγάλο κόπο στα τέλη Αυγούστου στο Κάιρο, αυτή η εκεχηρία να δρομολογήσει μια νέα πολιτική διαδικασία. Θα πω ότι την επόμενη εβδομάδα ε, θα είμαι σε μια ε, συνεδρίαση, σε ένα συνέδριο δωρητών ε, στο Κάιρο και ελπίζω να είναι εκεί και ο πρόεδρος Αμπάς για να συζητήσουμε συζητήσουμε και το πώς μπορούμε να ανοικοδομήσουμε πολιτικά τη Γάζα. Αυτό που θα ενδιαφέρει κυρίως είναι η, Ισραηλο, η Αραβο-Ισραηλινή διένεξη. Θα έχουμε λοιπόν μια ευρύτερη περιφερειακή προσέγγιση. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που είναι ωραίο στις ακροάσεις είναι ότι ε, μερικές φορές οι υποψήφοι εκπλήσονται για τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές ιεραρχούν τα θέματα. Ο κύριος Μελενσόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μελεντσόν, εάν προτιμάτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα γεγονότα που διαταράσσουν την παγκόσμια τάση της ανθρωπότητας. Ε, Εκπλήσουμε που δεν μιλήσατε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής ως πρώτο πρόβλημα στις σχέσεις των ε, εθνών. Πρώτη ε, και πρώτος λόγος των μελλοντικών μεταναστευτικών ροών. Τι θέση θα έχετε στη συζητήση στο Παρίσι όταν γίνει η συνοσκορυφής για το κλίμα. Το δεύτερο σημείο αφορά έναν τεράστιο παράγοντα διαταραχής, την πολύ ασταθή κατάσταση του δολαρίου ως διεθνές νόμισμα που διαταράσει όλες τις ε, σχέσεις του διεθνού συστήματος. Φέτος το καλοκαίρι έγινε ένα τεράστιο συμβάν. Ε, Ινδία, Βρασιλία, ε, Νότιο Αφρική κτλ. αποφάσισαν να δημιουργήσουν το αντίστοιχο του, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Δουνουτού μεταξύ τους. Και η, Ρωσία και η Κίνα αποφάσισαν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους να, ε, τα διεθνή τους ε, δικά τους νομίσματα. Αυτό που σημαίνει ότι δημιουργείται μία, μπαίνει το δολάριο σε μία έτσι πιο ασταθή θέση. Ευχαριστώ κύριε Μελενσού. Ανέφερα την κλιματική αλλαγή, που θεωρώ ότι είναι μία από τις πρώτες παγκόσμιες ε, προκλήσεις. Το είπα αυτό στην πρώτη μου παρέμβαση που έκανα στα αγγλικά. Πριν από λίγες εβδομάδες συμμετείχα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από το σημερινό Επίτροπο με τους Υπουργούς Εξωτερικών κάποιων κρατών μελών. Και νομίζω ότι η σύνθεση, για τη δική μου δουλειά τουλάχιστον, για το αξιωμά μου, αν το, με απόφαση επιβεβαιώσετε, μαζί με τον αρμόδιο επίτροπο, με τους υπουργούς εξωτερικών, με τους υπουργούς περιβάλλοντος, και το δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μας δίνουν και πληροφορίες αλλά και μας καταρτίζουν και διαμορφώνουν τις απόψεις μας. Στο εσωτερικό του ΟΗΕ όλη αυτή η συνάντηση, αυτός ο σχηματισμός θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο Παρίσι του χρόνου είπα ήδη ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε όλη την προεργασία που μπορούμε στη Λίμα το Δεκέμβριο. Εάν δεν κάνουμε στη Λίμα το Δεκέμβριο ένα τμήμα τη δουλειά, θα είναι πολύ προβληματική κατάσταση στο Παρίσι να τα καταφέρουμε. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε μία αποτυχία σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα ασφάλειας, διεθνούς ασφάλειας, όπως είπατε κι εσείς. Δεν είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα αυτό, το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Κύριος Μέσερης, ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία ε, Αριστήσα, είπατε εκπρόσωπε, εδώ είμαι. Χάρηκα που άκουσα ότι αναφερθήκατε ε, σε διαφοροποιημένη πολιτική ε, για τη γειτονία και την ανατολική και την νότια γειτονία. Και στην καλύτερη περίπτωση είναι μισή επιτυχία, ε, για να μην πω τίποτα χειρότερο αυτή η πολιτική. Άλλοι υποψήφοι επιτροποί περίπου ομόφωνα είπανε ότι είναι δική σας αρμοδιότητα η επαναχάραξη της στρατηγικής και θα σας ακολουθήσουν. Σε 5-6 μήνες από τώρα, ποιον θα πρέπει να ρωτήσουμε και να ζητήσουμε να έρθει να μας κάνει μια αναφορά στην Επιτροπή μας. Και μια πρακτική ερώτηση. Ε, η κυρία Ρεμπέκα Χάρμ, συμπρόεδρο μας, ε, ε, θα μάθατε ότι ανακηρύχθηκε persona non grata, ανεπιθύμητο πρόσωπο στη Ρωσία. Έχετε επίσημη πληροφόρηση γι' αυτό και τι σκοπεύετε να κάνετε για να το αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ για τις δύο ερωτήσεις. Ποιο θα ρωτήσετε για την χάραξη στρατηγική σε μένα. Ναι, σας το επιβεβαιώνω. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε μόνιμο αυτό βέβαια ξεκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, κλεισμένη μέσα στο γραφείο μου. Θεωρώ θετικό αυτό το μήνυμα, ότι θέλουμε ε, μια ε, ομαδική συνεργασία όλοι μας, αλλά βεβαίως χρειάζεται και καθοδήγηση και υπευθυνότητα ε, και αν με επιβεβαιώσετε, εγώ θα φέρω αυτή την ευθύνη. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ρεμπέκα, Harms, είμαι ενήμερη, όχι περισσότερο από εσά, μάλλον λιγότερο. Εσείς γνωρίζετε περισσότερα, καθώς δεν είμαι ε, σε θέση ε, αυτή τη στιγμή. Συμμερίζουμε απολύτως τα λεγόμενα του κυρίου Σούλτ, του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένας κατάλογος, ο οποίος ούτε δημόσιος είναι ούτε δικαιολογημένος τον προσώπο. Εάν με επιβεβαιώσετε θα ασχοληθώ βεβαίως και θα απευθυνθώ στις ρωσικές αρχές και θα ρωτήσω τι συνέβη. Και σε περίπτωση που δημοσίως ε, δικαιολογήσουν και αιτιολογήσουν αυτή την υπόθεση θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Α, να σας πω και το εξή εν παρόδο. Πιστεύω, έχω λίγο χρόνο ακόμα, ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία συγγνώμη, είναι κομβική σημασία. Και όποτε μπορώ να τη διευκολύνω είτε εγώ προσωπικά είτε οι υπηρεσίε μου για την πρόσβαση ή αποστολέ ευρωβουλευτών ε, σε χώρες που θέλουν να επισκέπτονται, όποτε μπορώ να το κάνω, να υπολογίζετε σε μένα ότι θα το πράξω. Από την άλλη θα σας ζητήσω και συντονισμό εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και για να καταλάβουμε καλύτερα ποιο είναι καλύτερα να είναι ο συνομιλητή, ποιο επισκεφ... θα επισκεφθούμε, χωρί να θέλουμε καθόλου να παρέμβουμε, αλλά για να υπάρχει μια συνεννόηση, γιατί υπάρχει και ο καρπός της κοινοβουλευτική δημοκρατίας ε, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, Με τρόπο όμω διαρθρωμένο και συντεταγμένο, για μένα βεβαίω, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πολύτιμα κυρία Λούνατσεκ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη. Στις ε, γραπτές σας απαντήσεις ε, είπατε ότι προτίθεστε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα χρησιμοποιήσετε ως πηξίδα στη δουλειά σας. Δύο ερωτήσεις λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλήσατε για τις γυναίκες, την θρησκευτική ελευθερία και θέλω να μας πείτε πώς θα ενδυναμώσετε τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων και των ε, σεξουαλικών μειονοτήτων στην Ευρώπη. Επίσης ε, υπάρχει το Αζερβαϊτζάν, μια χώρα όπου ασκείται πίεση του τελευταίους μήνε πολύ μεγαλύτερη πίεση κατά της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωση. Πώ σκοπεύετε λοιπόν να βελτιώσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. Και μια τελευταία ερώτηση που αφορά ε, στη θέση σα ε, της Ιταλίδα Υπουργού Εξωτερικών που ε, στηρίζει τον αγωγό South Stream. Θα ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο είναι κατά του South Stream γιατί δεν είναι ευρωπαϊκό έργο. Εσείς λοιπόν τι θα κάνετε ως Αντιπρόεδρος, γιατί θα ήθελα στο μέλλον να μείνετε ε, στη μνήμη των ανθρώπων, όχι ως η κυρία του South Stream, αλλά ως η κυρία του CFSP, του αγωγού CFSP της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ε, έχουμε ακόμα λιγάκι χρόνο να δουλέψουμε επ' αυτού. Κοιτάξτε, θα απαντήσω σε αυτό το θέμα πρώτα απ' όλα. Νομίζω λοιπόν ότι οι πολιτικές προϋποθέσεις για τον αγωγό South Stream, μπας περιπτώσει έτσι κι αλλιώς δεν είναι όριμες αυτή τη στιγμή. Και αυτό έχει σχέση με την Ουκρανία και με τι σχέσει μας με τη Ρωσία. Τα προγράμματα υποδομής πρέπει να έχουν μια σταθερή και σαφώς νομιμοποιημένη βάση. Όταν λοιπόν και εάν οι πολιτικές συνθήκες ομαλοποιηθούν με ένα μεγάλο εάν, τότε πιστεύω ότι οι τεχνικής φύσεως συζητήσεις μπορούν να ξαναξεκινήσουν και να δούμε τότε πια κατά πόσον θα μπορούμε, ε, θα είναι δυνατόν να καλύπτεται πλήρως η νομική βάση. Νομίζω ότι αυτή, αυτό ξεκαθαρίζει τη θέση μου. Όταν ήμουν εδώ ε, υπήρξε κάποια παρεξήγηση, νομίζω ε, κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν νομίζω ήταν βουλευτές, ε, με παρεξήγησαν. Εγώ είχα πει ότι ο νότιος αγωγός ε, θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας και ξέρετε ότι αυτός έχει σχέση με τον ΤΑΠ, ο νότιος διάδρομος που περνάει από το Αζερμπαϊτζάν. Δεν είχα πει για τον South Stream, ίσως ηχητικά να τον μπέρδεψαν. Επειδή λοιπόν επενδύουμε μεγάλα κονδύλια στην ενέργεια στο Αζερβαϊτζάν και το ξέρουν αυτό πάρα πολύ καλά ότι η δική τους εγωγή είναι καθοριστική σημασία και για τη δική μας τη διαφοροποίηση και για τις διαδρομές που θα ακολουθούν πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι και εκείνοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτικών ακτιβιστών. Όσον αφορά τώρα τις εθνοτικές ε, μειονότητες ε, και τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ και όπου μπορώ για να προστατεύσω τα δικαιώματά τους και θα το κάνω αυτό γιατί μακράδαν τα πεπισμένη, είναι στο DNA μου αν θέλετε, όχι επειδή πρέπει να το κάνω. Κυρίως όσον αφορά θέματα γενετήσιου προσανατολισμού σε κάποιες χώρες της Ευρώπης νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε αρκετά ακόμα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, ως Αντιπρόεδρος θα έχετε την ευθύνη του μέσου σταθερότητας και ειρήνης. Το μέσον αυτό τώρα στερείται 70 εκατομμύρια πληρωμές για φέτος και 60 για το 2015. Έτσι άμεσα μέτρα και επίγοντα ε, διαφύλαξη ειρήνης ε, εγκαταλείφθηκαν ή αναβλήθηκαν λόγω ελήψεως κονδυλίων. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι το μέσο σταθερότητας και ειρήνης έχει τη σωστή χρηματοδότηση. Και δεύτερη ερώτηση. Τι σημασία αποδίδεται ε, στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ΑΣΕΑΝ και τα κράτη-μέλη της ΑΣΕΑΝ, της Νότιο-Ατολικής Ασίας. Για τον προπολογισμό. Αν γίνω ύπατη εκπρόσωπος, θα συνεργαστώ με την Κρυσταλίνα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις, τη συνεργασία, ούτως ώστε άτυπα, ούτως ώστε να κάνουμε μια προσπάθεια. Ξέρω πολύ καλά την δέσμευση που έχει και μου δίνει αυτό ελπίδες ότι μαζί θα κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Ε, μάλιστα αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, το κάνουμε αμέσως. Και μετά αυτό που πρέπει να κάνουμε αργότερα θα το κάνουμε αργότερα. Γενικά υπάρχει πρόβλημα με τον προπολογισμό, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν αφορά μόνο αυτό το μέσο, το μέσο σταθερότητα και ειρήνη. Για τι φετινέ δεσμεύσει πληρωμών, οι δεσμεύσει πληρωμών που έχουμε πάνω σε αυτό το μέσο και σε όλε τι εξωτερικέ δράσει είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία μα. Και πιστεύω ότι η Κομισιόν το έχει απόλυτα το ξέρει αυτό πολύ καλά. Θα βασιστούμε και σε εσά για να βρούμε μια λογική λύση και για για να αναθεώρηση θα γίνει το 2016. Ίσως τότε μπορούμε να σκεφτούμε μαζί το θέμα, αν χρειάζεται να αναθεωρήσουμε κάτι στον προπολογισμό συνολικά. Και φυσικά θα έχουμε και μια άλλη ζήτηση για τον προπολογισμό για, για το 5% και τις περικοπές αυτές, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για τη σχέση με την ΑΖΕΑΝ, όπως ξέρετε, πριν από μερικές εβδομάδες ε, διορίστηκε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας το ΑΖΕΑΝ. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Είναι μία από τις στρατηγικές δουλειές που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια περιφερειοποίηση στην Ασία όπως και στη Λατινική Αμερική είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εάν δεν έχουμε μέσα ανάλογα με τις ανάγκες σε περιφερειακό επίπεδο, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Το να επενδύσουμε λοιπόν στις σχέσεις με την ΑΖΕΑΝ θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Fabio Castaldo. Ευχαριστώ, κύριε Μογκερίνη. Το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μιλάνε για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις διαστάσεις τη της εξωτερικής διάστασης. Είναι σημαντική αυτή η δέσμευση. Ξέρουμε ότι αυτές όμως οι ευρείες διατρανώσεις θυσιάζονται για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα σε εμπορικές σχέσεις. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά είναι επιλεκτική ως προς τις αρχές της. Ως μελλοντική είπατε εκπρόσωπος θα έχετε την ευθύνη για να συντονίσετε όλη την ομάδα των επιτρόπων που ασχολούνται με την εξωτερική δράση και επομένως τη δυνατότητα για να εξασφαλίσετε την συνεκτικότητα. Καλή τύχη. Μια και τα κράτη-μέλη. Ε, οι προσυπέγραψαν το πρωτόκολλο 13 για την κατάργηση του θανάτου, όπου για την κατάργηση της θανατικής ποινής, θεωρείται ότι είναι συμβατό το να διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία όπως το TTIP όπου ε, έχουμε χώρες που επιβάλλουν ακόμα την θανατική ποινή. Πώς ε, παντρεύονται αυτά τα δύο. Δύο ερωτήσεις. Ήταν αυτές. Δεν νομίζω. Σας ευχαριστώ για, την, ε, για το καλή τύχη που μου είπατε. Ε, Ελπίζω να με καταλάβατε στα Ιταλικά που το είπα, γιατί έτσι το λέμε εμείς. Για τη δουλειά που κάνουμε πάνω στην κατάρρηση θανατικής ποινής. Νομίζω ότι είναι το επισκεπτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτό το επισκεπτήριο. Η σύνδεση με την διαπραγμάτευση για την εμπορική συμφωνία ε, εδώ έχουμε να πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε διάφορα, έτσι. Είναι... Ίσως ο συσχετισμός λίγο προβληματικός που είπατε. Αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια καθολική απαγόρευση της θανατικής ποινή. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό μαζί με πολλούς ε, τέρους. Να ξεκινήσουμε με τις χώρες αυτές που δεν την κατάρρισαν αλλά έχουν οδηγηθεί σε μια αναστολή ούτω ώστε βήμα-βήμα να φτάσουμε στην πλήρη κατάργηση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να παίξει καθοριστικό ρόλο ε, σε αυτή τη μάχη, στο εσωτερικό του ΟΗΕ φυσικά. Και βεβαίω πρέπει να δημιουργήσουμε μια συμμαχία με τι οργανώσει κοινωνία των πολιτών που μπορούν να μα βοηθήσουν σε αυτή τη μάχη. Ε, μια και είσαστε Ιταλό, που με ρωτάτε, να σα δώσω ένα παράδειγμα από την Ιταλική ζωή. Δημιουργήσαμε, παραδείγματο χάρη, στην Ιταλία ως, ε, με δική μου πρωτοβουλία ως υπουργό ε, Εξωτερικών μια task force για την, για τη θανατική ποινή. Υπάρχει ένα νέο ψήφισμα για, την, ε, για το μορατόριο της θανατικής ποινής στο ΝΟΙΕ σε λίγο. Ε, έχουμε τρεις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολήθηκαν με αυτό. Δεν θέλω να τις αναφέρω για να μην κάνω διαφήμιση. Αλλά αν τα κρατημέλη, τα θεσμικά όργανα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι διάφορες οργανώσεις διάφορα κινήματα και διάφορε οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών μπορούν να δημιουργήσουν μια στρατηγική ούτω ώστε να προωθήσουν το μορατόριο και τελικά την κατάρριση τη αντική ποινή. Αυτό είναι ένα στόχο που τον θέλουμε και είμαι έτοιμη να δουλέψω από αυτού. Thank you, Chair. Madam, the member states... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να συστήσουν κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας ε, και μια κοινή αμυντική πολιτική. Ε, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της δικής σας της θητείας. Και πιστεύετε ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα έχει τον έλεγχο της δικής του εξωτερικής πολιτικής. Επίσης, μήπως αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα ουδετερότητας. Δεύτερη ερώτηση, πώς μπορεί να υπάρξει ε, αποτελεσματική εξωτερική πολιτική όταν υπάρχουν συνέχεια διαφωνίες στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη. Βλέπουμε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις, εσείς αυτές τις ε, καταδικάζετε και τι πιστεύετε σχετικά με την εθνική κυριαρχία του Γιβραλτάρ. Θα απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι το να διαμορφώνει κανείς ε, μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, ότι αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να παρετούνται από τη δική τους την ανεξάρτητη πολιτική, γιατί έτσι και αλλιώς και να τους το έλεγαν δεν θα το έκαναν. Αυτό μας βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιστούμε σε αυτό που απομένει. Αυτό λοιπόν που προσπαθώ να σας μεταφέρω είναι ότι είναι απαραίτητο για μας ε, να δημιουργήσουμε έτσι ένα αίσθημα κοινών συμφερόντων που να μπορούμε να τα προάγουμε, να τα υπερασπιστούμε με μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική όπου εντάσσονται οι διάφορες εθνικές πολιτικές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν θα αναλαμβάνουν ε, πρωτοβουλίες σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Μα δεν είμαι τόσο αφελής ε, να πιστεύω κάτι τέτοιο και δεν θα ήταν καν καλό κάτι τέτοιο. Γιατί πρέπει να υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κοινή κατεύθυνση, ένα κοινό όραμα και κάποιες κοινέ δράσεις για κοινά συμφέροντα και αξίες. Και επίσης είναι απαραίτητο να εργαστούμε όλοι μαζί για να τα διαμορφώσουμε αυτά. Όταν έφτασα στο θέμα της ιδιοκτησίας που ανέφερα στην αρχή με εισαγωγικά βέβαια, όταν φτάνουμε σε μια κρίση τότε δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική, έχουμε 28 εθνικές εξωτερικές πολιτικές και έναν κοινό παρονομαστή. Κάτι και αυτό, αλλά νομίζω ότι ε, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα και είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Το ζητούν αυτό οι πολίτες μας και οι πολίτες όμορων κρατών. Γι' αυτό σας λέω ότι θα είναι δύσκολο, αυτό θα είναι το πιο δύσκολο καθήκον που θα έχω να αντιμετωπίσω τα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και χρήσιμοι Ευρωπαίοι στους υπόλοιπους πολίτες και στους πολίτες του υπόλοιπου κόσμου, αν τελικά κατορθώσουμε να γραμματίσουμε πλήρως το ρόλο μας. Ε, κυρία Μογκερίνη, κυρία Προτινόμενη Επίτροπε, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή Πάνω από 15 εκατομμύρια παγκοσμίω ε, καταναλώνουν παράνομα οπιούχα που είναι μορφήνη, ηρωίνη και όπιο. Και ε, οι περισσότεροι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από την ηρωίνη και όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που αναγκάζονται ε, να έχουν θεραπεία ή να ζητούν για αυτά τα παράνομα ναρκωτικά ναρκωτικά. Η ηρωίνη δημιουργεί και οξέα και ε, ε, χρόνια προβλήματα, ε, C και AIDS λόγω της ενδοφλέβειας χρήσης. Ε, χιλιάδες είναι νεκροί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από τα θέματα υγείας, ε, αυτή η παράνομη βιομηχανία έχουν επηρεάζει και τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε πολλά μέρη του κόσμου και μάλιστα με χρηματοδότηση που δίνει σε αντάρτες σε ε, ε, περιοχές παραγωγής ιδιαίτερα στο Αφγανιστάν. Ερωτώ, εσείς πώς προτίθεστε να προστατεύετε τους πολίτες της Ευρώπης από αυτό το ε, επικίνδυνο πρόβλημα ναρκωτικών που στερεί τόσες ζωές και βλάπτει και την κοινωνία. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα ήταν χρήσιμο να συνεργαστούμε φανταστεί ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ομάδα. Γιατί ε, άπτονται διαφόρων δράσεων και διαφόρων τομέων πολιτικής και εσωτερικής και εξωτερικής. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο Αφγανιστάν. Ξεπλάγει που δεν αναφέρθηκε κανείς αυτό μέχρι τώρα και είναι ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη νέα αφγανική κυβέρνηση Σίγουρα τα τελευταία 13 χρόνια δεν ήταν ε, αποτελεσματική αντιμετώπιση. Βεβαίως είναι ένα θέμα κοινωνικής αποσταθεροποίησης, μάλλον είναι ε, πηγή αποσταθεροποίησης, είναι πηγή ε, χρηματοδότησης και θα πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε και όχι μόνο στο Αφγανιστάν, προφανώς και σε άλλα μέρη του κόσμου συμβαίνει αυτό. Βεβαίως λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι ένα τμήμα το χαρτοφυλακίου μου την επόμενη πενταετία αν αποφασίσετε να με επιβεβαιώσετε στη θέση αυτή. Ε, ο κύριος Εμρίκ Σοπράντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπάτη, ε, εκπρόσωπο, προτινόμενη είπατε. Πριν από λίγες μέρες ο Τζο Μπάιντεν, ε, Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ε, δήλωσε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει, και το τονίζω, επιβάλει, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε στους Ευρωπαίους, κυρώσει κατά της Ρωσίας. Ε, θυμούμε τα όσα είπατε για τη Ρωσία, σοφά λόγια και ισορροπημένα. Σήμερα άκουσα όμως ότι η προτεραιότητα θα ήταν η διατλαντική εταιρική σχέση, το ΝΑΤΟ, λογικές διεύρυνσεις προς Μολδαβία, Τουρκία, Αζερβαϊτζάν, Γεωργία. Κυρία προτινόμενη είπατε πρόσωπε, νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι εδώ θα ήταν πιο ήσυχοι αν τους καθησυχάζατε και τους επιβεβαιώνατε ότι θα είστε πρόσωπος της Ευρώπης ε, ανεξάρτητης δύναμης και όχι ενός διατλαντικού συνασπισμού που θα κυριαρχούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Βεβαίως και θα είμαι. Ε, αν με επιβεβαιώσετε στη θέση αυτή και κατά τα άλλα. Ε, μ' αρέσει η προσφώνηση στα γαλλικά από ότι στα αγγλικά. Εγώ δεν μίλησα ποτέ για να το διευκρινίσω ε, για διεύρυνση προς τις χώρες αυτές. Είπα ότι η πολιτική διεύρυνση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας προς το παρόν ήταν επιτυχής και νομίζω και στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτό. Κατά τα άλλα έχουμε καλές ε, σχέσεις εταιρικές και γειτονίας και θα πρέπει να ε, δούμε αναχώρα ε, την κατάσταση. Διάβασα κι εγώ τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος ε, Biden και μάλλον εξεπλάγεν από τα λόγια του αυτά. Γιατί συνεργαστήκαμε όχι με τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν, αλλά κατά κύριο λόγο οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, αλλά και σε ένα διάλογο όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με άλλες χώρες ε, που είχαν την ίδια στάση και επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία. Ε, βλέπε Ιαπωνία, ε, Καναδάς κτλ. Συνεργαστήκαμε λοιπόν για να συντονιστούμε για μια διεθνή και θα έλεγα παγκόσμια προσπάθεια. Μπορώ να σας πω όμως από την άμεση εμπειρία που έχω αποκομίσει ως υπουργό στην Ιταλική κυβέρνηση ότι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ήταν ποτέ εύκολες, αλλά είναι πάντα αυτόνομες, ανεξάρτητες, βασίζονται στην ενδοευρωπαϊκή συζήτηση και με εκπλήσει το γεγονός ότι υποχρεώνουμε να το τονίσω αυτό. Για μένα αυτό είναι προφανές και αυτονόητο μεταξύ μας. Μόνο έτσι νοείται η λήψη των αποφάσεων στην Ευρώπη. Ήταν δύσκολη η απόφαση αυτή να ληφθεί για πολλές χώρες, πολλές κυβερνήσεις, αλλά ανέκαθεν ήταν μια κοινή ε, απόφαση και ένας κοινός προβληματισμός. Και επαναλαμβάνω, ήταν πολύτιμη η αξία της ενότητας της Ευρώπης σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις αρχικές σας παρατηρήσεις κάνετε μια αναφορά στην Ασία. Συμφωνείτε ότι οι έντονες σχέσεις με την Ασία είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί η Ασία έχει το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού και ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου ΑΕΠ. Τα νούμερα αυτά θα αυξηθούν μάλιστα δεδομένων των οικονομιών στην περιοχή που κρατάνε τα σημερινά επίπεδα ανάπτυξης. Επίσης η Ασία όμως είναι εστία πολλών ε, θεάτρων πολέμου και μπορούν αυτές οι σειράξεις να απλωθούν προς τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα να θέσω λοιπόν τρία ερωτήματα. Καταρχάς, έχουμε μια νέα κυβέρνηση στην Ινδία, τον Πρωθυπουργό Μόντι. Και δεν είναι πουθενά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ συναντάτε με την Ιαπωνία, το, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους πρωθυπουργούς και τους πρόεδρους των χωρών αυτών. Και αυτές είναι οι προτεραιότητες τους. Πέρασε μια δεκαετία από τότε που ξεκίνησε η στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας, που όμως δεν έδωσε καθόλου καρπούς. Μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε να συνεχίσω. Όχι. Οι σχέσεις με την Ασία θα είναι στρατηγικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόκληση είναι να δείξουμε στην Ασία ότι και για αυτούς η σχέση μαζί μας είναι στρατηγική σημασία. Γιατί υπάρχει τόσος ανταγωνισμός εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλή προσπάθεια, κοινή προσπάθεια και να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Γιατί η Ασία είναι μια τέτοια ήπειρος που η κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο μπορούμε εμείς να, πρέπει εμείς να γίνουμε σημαντικοί για αυτούς. Όπως και αυτή είναι σημαντική για μας, για την Ινδία πιο συγκεκριμένα τώρα. Πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση στην Ινδία η οποία προσπαθεί να ανοιχτεί και να δημιουργήσει δεσμούς με τον υπόλοιπο κόσμο, είναι μια ευκαιρία. Τώρα που έχουμε και μια νέα ηγεσία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να βράξουμε αυτή την ευκαιρία, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τους δεσμούς. Ε, Κύριε Σπανιό. Κυρία υποψήφια, είπατε εκπρόσωποι, τα σύνορα ε, Μαρόκου-Αλγερίας είναι κλειστά εδώ και δεκαετίας. Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες δεν βελτιώνεται. Δεν υπάρχει καμία περιφερειακή συνεργασία στο Μαγκρέμπ. Κάτι που θα ήταν θετικό και για τους πληθυσμούς της Νότιας Μεσογείου, αλλά και στην Ευρώπη, χάρη σε νέες προ... προοπτικές εταιρικής σχέσης. Τα αποτελέσματα είναι πικρά. Το Μαγκρέμπ είναι ένα μπλοκ που είναι πολύ λίγο ολοκληρωμένο. Εμείς κάνουμε προσπάθειες ε, για συνεργασία. Ε, επίσης, ε, η Σαχάρα είναι τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύσει την επίλυση αυτών των διαφορών και να μπορέσει να βοηθήσει στην συμφιλίωση του Μαρόκου και της Αλγερίας. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρώπη για την ε, δημιουργία της Ένωσης του Μαγκρέπ που θα μπορούσε να δώσει ένα όραμα ειρήνης. Τέλος, τι δράσεις ε, προβλέπετε για να παίξει ένα σημαντικό ρόλο η Ευρώπη στο Μαγκρέπ τη στιγμή όπου και διακόπτει ο Πρόεδρος. Φινίτο δυστυχώς. Δεν φταίω εγώ, λέει η κυρία Μογκερίνη. Γερμανική ευελιξία είναι αυτή. Sorry. Συγγνώμη κύριε Μπρόκ γι' αυτό. Συγγνώμη πρόεδρε. Ναι, ναι, ξέρω, δεν ήταν πολύ διπλωματικό αυτό που είπα και δεν είμαι διπλωμάτης. Εστιάζουμε στο αποτέλεσμα, εντάξει. Μπορώ να τελειώσω και εγώ, λέει ο κύριος Πανιού. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Και ζητώ συγγνώμη για τον αστερισμό. Είναι παράδοξο ότι η λιγότερο ολοκληρωμένη περιοχή είναι η περιοχή του Μαγκρέμπ. Και όμως εκεί χρειαζόμαστε την περιφερειακή ολοκλήρωση. Όταν βλέπουμε τη δουλειά που γίνεται στη Λιβύη με τις γειτονικέ χώρες, μέσα σε ένα δύσκολο σχήμα, αλλά απαραίτητο, 5 συν 5, όπως σας είπα και προηγουμένως, βλέπουμε ότι αυτό δίνει καρπούς. Φυσικά υπάρχουν διμερεί προβλήματα. Μαρόκο, Αλγερίας. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρώπη. Καταρχάς, είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για μια πολιτική λύση, ευρεία, και βιώσιμη του, της σύγκρουσης στη Δυτική Σαχάρα, να χρησιμοποιήσει τις περιφερειακές μορφές διαλόγου που έχουμε για να συνεργαστούμε, γιατί έχουμε μια πρακτική έτσι, κοινής δουλειάς και αυτό διευκολύνει τα πράγματα και να δουλέψουμε και στις διμερείς σχέσεις που έχουμε με το Μαρόκο και την Αλγερία την άλλη, για να περάσουμε το μήνυμα ότι έχει νόημα να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Χωρί μια περιφερειακή προσπάθεια, μια πραγματική περιφερειακή προσπάθεια, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε πραγματικές λύσεις της κρίσης στη Λιβύη. Χρειαζόμαστε χρόνο για να δουλέψουμε, για να ανταλλάξουμε ιδέες και είμαι πεπισμένη ότι θα είναι το πρώτο θέμα τους επόμενους μήνες τα επόμενα χρόνια για την ε, ασφάλεια, τη δική μας και τη δική τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι ότι ακόμα δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως τη συνθήκη της Λισαβόνας και γι' αυτό θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Πώς θέλετε και πώς μπορείτε να πετύχετε τα κράτη-μέλη να επιτύχουν, δηλαδή να έχουν ε, καλύτερη χρήση και εκμετάλλευση της ε, συνεργασίας. Επίσης, ε, πώς θα προσπαθήσετε να εκμεταλλευτείτε τη συνθήκη της Λισαβόνας κυρίω για θέματα εξοπλισμών και τι θα κάνετε συγκεκριμένα έτσι ώστε να διατηρήσετε διατηρήσετε και να σταθεροποιήσετε την ευρωπαϊκή βάση των εξαπλισμών. Επίσης, πώς θα μπορέσετε να διασφαλίσετε ότι ε, θα καλυφθούν ε, τα κενά που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως ε, τα θέματα που προσφέρει ο οργανισμός. Στην Αφρική, Εκεί στο μέλλον ε, θα υπάρχει το African Peace Facility. Τι θα κάνετε με αυτό. Και μία άλλη ερώτηση. Τη στρατηγική ασφάλεια της Ευρώπης σκοπεύετε να την ε, χρησιμοποιήσετε και για την κατάρτιση μιας λευκής βίβλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας τις ερωτήσεις. Ξεκινάω από την διατρομένη συνεργασία. Όπως θα έχετε διαπιστώσει, αυτό υπάρχει στις γραπτές μου απαντήσεις και σκοπεύω τα επόμενα πέντε χρόνια να τα εκμεταλλευτώ για να δω αν θα υπάρχουν οι πολιτικές συνθήκες για να ε, προωθήσω αυτό το θέμα, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες τότε πράγματι θα είναι καθήκον μου να εξετάσω το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον οργανισμό άμυνας, ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι υπάρχει εκεί ένα τεράστιο δυναμικό και εγώ ε, θέλω να συνεργαστώ με τους ε, υπουργούς άμυνας που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου θα προείσταμε. Να έχουμε λοιπόν μια κοινή προσέγγιση. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και τους πρώτους μήνες από την ανάληψη της θητείας μου. Ε, έχουμε Συμβουλίο Υπουργών Άμυνας τον Νοέμβρη. Θα υπάρξουν ε, κάποιες αλλαγές ε, στις αρχές του έτους. Αυτό είναι ένα από τα θέματα όπου σήμερα ε, δεν μπορώ να σα δώσω κάποιες συγκεκριμένε απαντήσεις, δεν έχω βέβαια και το χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι στι πρώτε μου προτεραιότητε. Και κάτι που θα κάνω διαφορετικά από το παρελθόν είναι ότι ε, θα εξηγήσω ακριβώ το ρόλο μα σε θέματα Άμυνα. Τώρα για την ε, στρατηγική ασφάλεια. Έχω πει ότι αυτή τη στιγμή δεν έρχομαι σε εσά με σαφείς απόψεις για το κατά πόσον ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή μια διαδικασία όπως είναι η Λευκή Βίβλος. Αν ε, πρόκειται απλά για στρατηγικές σκέψεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με μία ευελιξία. Κοιτάξτε, δεν έχω ακριβώς τον τύπο, αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ε, στρατηγική σκέψη, κοινή στρατηγική σκέψη. Κύριος Ποστινάρου, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη ε, Φεντερίκα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλωσορίζει πάρα πολύ την προσήλωσή σας για τη στρατηγική επαναχάραξη ε, του συντονισμού των ε, παγκοσμίων πολιτικών και είμαι βέβαιος και πεπισμένος ότι το Κοινοβούλιο θα σας υποστηρίξει απολύτως. Ε, η κρίση έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα ε, και αυτό δημιουργεί προβλήματα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τον εφοδιασμό σε ενέργεια. Μετά το περασμένο θέρος, οι πιο σοβαρές κρίσεις ε, ήταν ε, την ε, ε, σύγκρουση Ισραηλινών Παλαιστινίων. Θα πάτε στο Κάιρο πιθανόν στην διάσκεψη των δωριών, ρητών. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι γι' αυτό ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να είναι ε, πλέον πληρωτής αλλά παίκτη, όχι payer αλλά player. Ωραία. Ποια θα είναι η στρατηγική σας για τις ενευτικές συνομιλίες και για την επιτέλους επίτευξη ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Σε δύο λεπτά να σας τα πω αυτά. Πρώτον, θα πρέπει να είμαστε παρόντες διότι για πρώτη φορά στα χρονικά υπάρχει και ανάγκη και αίτημα από όλες τις πλευρές να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με διαφορετικό τρόπο σε κάθε πλευρά, αλλά και ε, μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών και των περιφερειακών δυνάμεων. Μας το ζητούν και οι Αιγύπτιοι και οι Λυποί. Ε, θα έχουμε ένα κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση. Νομίζω ότι οι συνομιλίες έχουν πάρει πάρα πολύ χρόνο. Αν έχουμε την πολιτική βούληση να ε, εξευρεθεί μια πολιτική λύση, πρέπει να προχωρήσουμε. Η τεχνική λύση βρίσκεται. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση και η πολιτική καθοδήγηση και στους δύο τομείς και εντός των δύο. Ο ρόλος μας λοιπόν θα πρέπει να είναι να ασκήσουμε πολιτική πίεση Είμαστε πολύ μεγάλη χορηγή εκεί, οπότε έχουμε τη δυνατότητα πίεσης και ε, άσκησης ε, αυτής και παροχή κινήτρων. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική βούληση στην ε, περιοχή. Πρώτον, θα πρέπει να επιτραπεί στην Παλαιστινιακή Αρχή να κυβερνάει στην Γάζα. Γάζα. Άκουσα θετικά νέα, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, η κυβέρνηση συνοχής της Παλαιστινιακής Αρχής ε, για πρώτη φορά συνεδριάζει στη Γάζα την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν απατώμε. Θα πρέπει ε, να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ ε, μεγάλη δυνατότητα έχει η Ένωση να βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή για μεταρρυθμίσεις, για ελέγχους, να γίνεται σωστά η ανοικοδόμηση, γιατί θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις Ισραηλινές ανησυχίες ότι η ανοικοδόμηση να είναι ουσιαστική ανοικοδόμηση και όχι ε, Αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε να θέσουμε στη διάθεση ε, της υπόθεσης με υποστήριξη των πρακτικών συμφωνιών είναι δεδομένα. Αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζεται πολιτική βούληση, διότι η κρίση του καλοκαιριού τι λέει στην κοινή γνώμη της κάθε πλευράς ότι δεν υπάρχει ε, περίπτωση να επανέλθουμε στο status quo. Ο κύριο Μιγιάν Μουν. ευχαριστώ. Κυρία Μογερίνη, οι σημαντικότερε στρατηγικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, αυτέ που έχει με τι ΗΠΑ. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, όπω είπατε, σε ένα διεθνέ πλαίσιο τόσο δύσκολο. Αυτή η σχέση με τι ΗΠΑ θα είναι ακόμα πιο ε, ισχυρή εάν ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις ε, ε, τη συμφωνία TTIP. Και επίσης, τι θα κάνετε έτσι ώστε στην Ουάσιγκτον να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο οικονομική δύναμη και εμπορική Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολιτικός ε, πρωταγωνιστής. Χαίρομαι πολύ για αυτά που είπατε για τη Λατινική Αμερική. Είναι μια περιοχή που είναι φιλόδοξη στην ολοκληρωσή της, διεθνή παρουσία, ε, που αναβαθμίζεται. Οι περισσότερες είναι χώρες με δημοκρατικές αρχές και αξίες και διεισδύει πολύ έντονα εκεί η Κίνα. Τον Ιούνιο στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες τι θα κάνετε για να αναζωογονηθεί αυτή η σχέση. Και τέλος χαίρομαι για αυτό που είπατε για τη Μεσόγειο, για τις χώρες που είναι γειτονικέ μας και τόσο σημαντικές για μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες είναι στρατηγική, το είπα, αλλά και πολύ σημαντική από πολιτικής πλευράς. Πρέπει να ζήσουμε 100% το δυναμικό της διατλαντικής μας σχέσης. Πριν από λίγο καιρό, κάνα χρόνο, ίσως 1,5 χρόνο, στην Ευρώπη ξέσπασε πανικός. για το γεγονός ότι θεωρήσαμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, μας εγκαταλείπουν και στρέφονται προς την Ασία. Και μετά από ένα χρόνο μιλάμε για την ενδυνάμωση της σχέσης μας, ε, για την ενδυνάμωση της διατλαντικής σχέσης. Σημαντικό και για τη διάσταση της ασφάλειας. Είναι σημαντικό να οριμάσει αυτή η σχέση. Όπως δεν είναι σωστό να πανικοβληθούμε, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τρέχονταν και προς τον ειρηνικό, ούτε τώρα πρέπει να ξεχάσουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί με τους Αμερικανούς στον κόσμο. Εγώ έτσι το βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα μαζί. Μαζί μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τρίτες χώρες, να αντιμετωπίσουν κάποιες από τις παγκόσμιες απειλές, παραδείγματος χάρη την κλιματική αλλαγή, τις μεταναστευτικές ροές, τι δουλειά πρέπει να κάνουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε πολλού άλλου τομεί όπου η εταιρική σχέση είναι σημαντική. Κοινέ προσπάθειε που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τον έμπολα, Φερρυπίν. Υπάρχουν πολλέ ίδιε απόψει και λόγοι για να δουλέψουμε με του Αμερικάνου για τι διαπραγματεύσει για το TTIP. Δίδεται μεγάλη προσοχή από εσά, το ξέρω. Είμαι πεπισμένη ότι μπορεί να είναι στρατηγικό εργαλείο Εξωτερική πολιτική, όχι μόνο ε, εμπορική πολιτική. Ξέρω επίσης ότι υπάρχει μια κατανοητή αγωνία για το αν θα είναι καλή συμφωνία. Νομίζω ότι έχουμε όλο το χρόνο για να διαπραγματευτούμε το TTIP με τέτοιο τρόπο για να φτάσουμε σε μια καλή συμφωνία. Ο πρόεδρος Γιούνκερ, αυτά που είπε στο, στο Στρασβούργο, στο, στην Ολομέλεια, εγώ δεν θέλω μια οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά θέλω μια καλή συμφωνία με συγκεκριμένε προποθέσει, είπε ο Γιούνκερ. Και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο βεβαίω ε, το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται 100% για όλα αυτά τα θέματα. Η κυρία Αλιό Μαρή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μαγκερίνη. Για τη συνεργασία με τις χώρες του κόλπου. Έχουμε την ε, συνεργασία κατά τον Ταέσο. Είναι σημαντικό για τη στρατηγική. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε το δυναμικό αυτών των στρατηγικών εταίρων στο τομέα της ε, ασφάλειας και της άμυνας και στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις σχέσεις μαζί μας. Και τι δράσεις ε, προβλέπετε. Επίσης, το Συμβούλιο Συνεργασίας είναι για μας εμπορικός εταίρος σημαντικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διμερείς σχέσεις με τις χώρες του κόλπου χάρη στην Συμφωνία Συνεργασίας του 88 και από το 2008 οι διαπραγματεύσεις για την, ε, τις ελεύθερες συναλλαχές παρενέβησαν. Πώς θα επανεκκινήσει αυτή η συνεργασία. Θα πάρει νέα ορμή και στα πλαίσια της ε, ε, ενεργειακής κρίσης της Ευρώπης. Πώς αξιολογείται τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών. Λοιπόν, δεν θα, δεν θα μιλούσα για στρατιωτική συμμαχία και συνασπισμό των χωρών αυτών. Θα την ε, ονόμαζα συνεργασία, συνασπισμό. Γιατί δεν είναι μόνο ε, στρατιωτικός. Υπάρχουν χώρες ε, που συμμετέχουν στο συνασπισμό και κάνουν, έχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά και χώρες που συμμετέχουν στι στρατιωτικές επιχείρησεις δεν συμμετέχουν στο ε, συνασπισμό. Υπάρχει ε, ο υπεύθυνο για να συντονίσει τις προσπάθειες του, του συνασπισμού, ο οποίος, με τον οποίο συνομίλησα. Και συμφωνεί μαζί μου ότι πρέπει να έχουμε όχι μόνο αποτελεσματικές στρατιωτικές δράσεις, αλλά και δράσεις άλλου τύπου. Για το επίπεδο χρηματοδότησης, για το οικονομικό θέμα, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η συμμετοχή των χωρών του κόλπου είναι πολύ σημαντική. Και έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τη δυναμική στην περιοχή. Και δεν είναι καθόλου εύκολο, έτσι. Και ήδη βλέπουμε πόσο περίπλοκο είναι. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετικά συμφέροντα. και κινείται προ διαφορετική κατεύθυνση από του υπόλοιπου, ανάλογα με τα συμφέροντά του. Όμω, η συμμετοχή των χωρών στο συνασπισμό αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα αυτό, το πρόβλημα του Ισλαμικού κράτου είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χώρε τη περιοχή. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν έχουμε να κάνουμε ένα Ιρακ Δεν είναι μια σύγκρουση πολιτισμών αυτή που συμβαίνει εκεί. Δεν αντιπαρατίθονται θρησκείες και πολιτισμοί. Όλοι μαζί είμαστε, όλοι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια τρομοκρατική οργάνωση. Για την επανεκκίνηση της εταιρικής σχέσης με τις χώρες του κόλπου είχα την ευκαιρία να αντικαταστήσω την Καθρινάστον ως υπουργό Τη Ιταλική προεδρία, δηλαδή Υπουργό Εξωτερικών, στη συνάντηση που είχαμε με τις χώρες του κόλπου και αρχίσαμε να συζητάμε πώ θα δώσουμε νέα πνοή στην εταιρική σχέση και σε οικονομικό και σε εμπορικό επίπεδο. Λοιπόν, ε, τελευταίες ε, δύο ερωτήσει, παρακαλώ. Ε, Τούνα Κέλαμ. Κυρία υποψήφιε επίτροπε, αυτό που με εντυπωσίασε είναι ε, θα θελήσετε να εφαρμόσετε σωστή εξωτερική πολιτική, αλλά δεν πείσατε ακόμα πώς θα σταματήσετε, πώς θα αναχαιτήσετε τον κύριο Πούτιν. Ε, ο, η Μόσχα είναι εκείνη που καθορίζει τα θέματα και εμείς ακολουθούμε, απλώς αντιδρούμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω, δεν πιστεύετε κι εσείς ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να καταδικάσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της ρωσικής επιθετικότητας. Υπάρχει αυτό το σκάνδαλο της ε, στρατιωτικής επέμβασης ε, και αυτό το δόγμα έχει οδηγήσει στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά την Ουκρανία, πώς είναι δυνατόν να αρνείται κανείς όπλα σε μία φίλη χώρα που δέχεται επίθεση Εάν αυτό δεν σημαίνει ότι ξεπερνιέται η κόκκινη γραμμή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τότε ποια είναι η κόκκινη γραμμή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές από όλους μας, από μας Ήδη ευθύ εξ αρχής, από τότε που ξέσπασε η κρίση, όλοι ξέρουμε ποιος φέρει την ευθύνη και πόσο επικίνδυνο είναι όχι μόνο για τη δική μας την Ήπειρο, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο το να αλλάζουν σύνορα με τη βία. Και νομίζω ότι αυτή είναι η βάση όλων των αποφάσεων που λάβαμε τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία, ανάμεσά μας τουλάχιστον, ότι όποια και είναι η πολιτική μας οικογένεια ή το κράτος μέλος ή η προσωπική μας άποψη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το να αλλάζει κανείς τα σύνορα με τη βία, να κάνει προσάρτηση μιας χώρας, να εγκαθιστά στρατεύματα σε μια ξένη χώρα, αυτό σαφώς και σημαίνει παραβίαση των διεθνών αρχών επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει και που αποτελούν τη βάση της δουλειάς μας. Το θέμα είναι πώς όλα αυτά μπορούν να γίνουν αποτελεσματικά για να αναχαιτιστεί ο Πούτιν. Και νομίζω σε αυτό το ερώτημα θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε μια ενδελεχή συζήτηση. Καταρχήν με τους φίλους μας από την Ουκρανία. Το δικό μου το σημείο αναφοράς είναι να δουλέψουμε με τους Ουκρανούς, γιατί σε τελική ανάλυση εκείνη είναι Εκείνοι ζουν στην περιοχή, αυτοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τη σύγκρουση στα εδάφη τους και με αυτούς τελικά προσπαθούμε να καταρτήσουμε μια στρατηγική για να αναχαιτήσουμε την κατάσταση. Έχουμε υιοθετήσει κυρώσεις. Τώρα, κατά πόσον οι κυρώσεις ήταν αποτελεσματικές στην ρωσική οικονομία, ναι, ήταν. Εγώ νομίζω ότι η ρωσική οικονομία αρχίζει να υποφέρει ουσιαστικά από τις κυρώσεις. Αν λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον επηρεάσαμε τη ρωσική οικονομία, η απάντηση είναι ναι. Αν επηρεάσαμε τις πολιτικές αποφάσεις της Ρωσίας, εκεί εξακολουθεί να υπάρχει ένα ερωτηματικό. Και οι Ουκρανοί έχουν κάποιο ερωτηματικό, γιατί τώρα αρχίζουν να λένε ότι πρέπει να εργαστούμε για να βρούμε μια πολιτική λύση. Άρα δηλαδή εγώ πιστεύω αυτό που έχει ε, σημασία είναι να στηρίξουμε τον Ουκρανό πρόεδρο και να συμφωνήσουμε μαζί του τα βήματα που θα κάνουμε. Ο κύριος Πέτρελα. Καλησπέρα σας κυρία Προτινόμενη Επίτροπε. Ως τελευταίος ομιλητής ε, θα σας ευχηθώ να μην είστε μόνο ύπατοι αλλά και ισχυροτάτοι Αντιπρόεδρος. Αναφερθήκατε στα Δυτικά Βαλκάνια. Ποιες θα είναι οι δικές σας προτεραιότητες σε συνεργασία με τον Επίτροπο Χάν για να αλλάξει η αρκετά ασύμετρη εικόνα των Βαλκανικών κρατών ως προς την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Συμφωνείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη όταν είναι έτοιμη μια υποψήφια χώρα. Πώς βλέπετε την Τουρκία σε αυτό το πλαίσιο. Ήδη αναφερθήκατε στην Ινδία. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο παραπάνω ότι θα κάνετε για να εμβαθύνετε τη συνεργασία με την Ινδία που για μένα είναι όλο και πιο σημαντικό στρατηγικό εταίρος για την Ένωση. Βέβαια την ίδια ερώτηση έχω και για την ε, Ιαπωνία. Ευχαριστώ. Για τα Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπει τελευταία ερώτηση να μιλήσω για τα Βαλκάνια. Νομίζω δεν θα ήταν δίκαιο να έχουμε μία προτεραιότητα εκεί, διότι η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής πορείας όλων των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων είναι η περιφερειακή διάσταση και οι αλληλεπιδράσεις και οι δεσμοί που έχουν μεταξύ τους. Είναι πιο εύκολο να πάει κανείς ε, από τις πρωτεύουσες στη Φραγκφούρτη ή στη Βιέννα, ή στη Βιέννη, συγγνώμη, ε, παρά από τη μία πρωτεύουσα στην άλλη. Ε, είναι και ένα θέμα διασυνδέσεων μεταξύ τους δεν είναι ολοκληρωμένη η ε, περιφέρεια εκεί, δεν υπάρχει αυτή η περιφερειακή ολοκλήρωση. Ε, είναι πολλές οι προτεραιότητες λοιπόν, αλλά οι καταστάσεις πολύ διαφορετικές και θα πρέπει να τις δούμε πολύ διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει μόνο ένα προτεραιότητα είναι η Βοσνία Ζεγοβίνη. Μετά τις εκλογές να ε, εφαρμοστεί το σύμφωνο για την ανάπτυξη και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Οι συνομιλίες Σερβίας, Κωσόβου επίσης. Συνεχίζονται σε επίπεδο τεχνικό, αλλά θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο αυτή τη στιγμή κυβέρνηση στην ε, Πρίστινα. Η Αλβανία έχει μοναδική ευκαιρία για τις μεταρρυθμίσεις. Το Μαυροβούνιο επίσης πρώτο-πρώτο στον κατάλογο. Και για τη Φυρό το θέμα της ονομασίας έχει να κάνει με πολιτική βούληση. Θα πρέπει να βρεθεί πολιτική βούληση για να επιληθεί. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει καμία χώρα. Για την Τουρκία σας ρώτησα. Ναι, ναι, αλλά εγώ μιλώ για τα Βαλκάνια. Για την Τουρκία μίλησα προηγουμένως και στην εισαγωγή μου. Ότι βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, και προς την Τουρκία την διεύρυνση. Ε, να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε, έτοιμη όταν είναι έτοιμες οι χώρες. Από κοινού Εκείνη είναι η πραγματική πρόκληση να ε, αποδώσει αυτή η πολιτική προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Δεν θέλουμε να έχουμε ε, έτσι μια πατεναλιστική προσέγγιση και να τους υπαγορεύουμε οτιδήποτε. Θα πρέπει από κοινού να είμαστε έτοιμοι την ίδια στιγμή.